Um, Καλησπέρα σε όλους σας εδώ στις Βρυξέλλες σήμερα το απόγευμα. Είναι η τελευταία μας συνεδρίαση αυτή για το 2012. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στον Πάνο έχει γενέθλια, χρόνια πολλά πάνω. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα, είναι ο επικεφαλής του τμήματός μας. Να ζήσει. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου τώρα. Θα το ξέρετε βέβαια, αλλά το λέω και για αυτούς που μας ακούνε στο διαδίκτυο. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Δεν θα ψηφίσουμε την έκθεση Τύρνεν για την οδηγία όσον αφορά τους εργαζόμενους για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα όλοι οι συγητές και όδες οι συγητές θεωρούν ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να καταλήξουμε σε έναν καλό συμβιβασμό. Δεν έχω αντίρρηση και εγώ. Πρόκειται για την απόσπαση εργαζομένων. Έκθεση της Emily Τούρνεν. Οπότε καλύτερα είναι να περιμένουμε για να βελτιώσουμε την ε, πρότασή μας. Γι' αυτό λοιπόν και δεν θα την ψηφίσουμε. Και ούτε είναι και στην ημερήσια διάταξη σήμερα το απόγευμα προς συζήτηση. Αυτό που θα κάνουμε ανταυτού όμω σήμερα το απόγευμα είναι ότι θα συζητήσουμε περισσότερο την έκθεση του κ. Ραμών για το δικό του θέμα που έχει να κάνει με τις υπηρεσίες και την ανταγωνιστική πολιτική, επίσης για την πολιτική ανταγωνισμού, την έκθεση ΣΦΑΜ θα συζητήσουμε. Στις 16.45 ε, θα αρχίσουμε τη συζήτηση. Συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη με τις αλλαγές αυτές. Ευχαριστώ. πρέπει να ξέρετε. Αύριο το πρωί προβλέπετε φωτογράφηση, δηλαδή πριν αρχίσει η συνεδρία των συντονιστών, αύριο το πρωί να είσαστε εδώ για να έχουμε μια οικογενειακή φωτογραφία. Επίσης, να ξέρετε ότι υπάρχει εδώ πέρα το newsletter μας. Υπάρχει αντίγραφο το οποίο μιλάει για τις εργασίες μας. Είναι και το χριστουγεννιάτικο τεύχος, βγήκε και την ημέρα που έχει τα γενέθλιά του ο Πάνος. Πολύ συχνά ε, μας ρωτάτε για τις διαπραγματεύσεις και τους τριμερείς διαλόγους. Οποιοδήποτε πάντως κοιτάξει και στο διαδίκτυο και εδώ στο newsletter θα δει πληροφορίες για αυτά. Επίσης να σας πω ότι από την τελευταία φορά που βρεθήκαμε μέχρι σήμερα έχει υπάρξει συμφωνία με το Συμβούλιο για τις διαδικασίες ε, ADR και ADR. Να ξέρετε ότι υπάρχει λοιπόν αυτή η συμφωνία. Είναι για τις συλλογικές προσφυγές και Και, και τα αναλλακτικά μέσα διευθέτησης διαφορών. Το Συμβούλιο μου επιβεβαιώνει ότι εφόσον ε, συμφωνήσει στην πρώτη ανάγνωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τότε τη θέση αυτή θα την εγκρίνει και το Συμβούλιο. Αυτό λοιπόν είναι το συμπέρασμα της όλης διαδικασίας. Πάντως να ξέρετε ότι αύριο θα σας δοθεί ευκαιρία να συμφωνήσετε και επίσημα και ευκαιρία να ευχαριστήσω και τον κύριο Γκρέκ αλλά και τους σκιώδεις συζητητές. Αύριο θα είναι εδώ όλοι και μετά. Το Φεβρουάριο νομίζω θα καταφέρουμε να το πάμε στην Ολομέλεια το θέμα αυτό για να ψηφιστεί εκεί. Οπότε είναι το δεύτερο πράγμα για την ολοκλήρωση της ενίας αγοράς που ολοκληρώνουμε. Και Τώρα για το θέμα του RPR. Να ξέρετε ότι βρισκόμαστε σε τριμερή διάλογο την πέμπτη το πρωί. Πολύ σημαντικό θέμα που ολοκληρώνεται επίσης. Τώρα πάμε στην έκθεση του κύριου Μπαλτασάρε. Προηγουμένως όμως θέλω να σας ενημερώσω ότι η κυρία Ρέντινγκ ζήτησε να βρεθεί μαζί μου. Αποφασίσαμε στις 4 παρατέταρτο. Ο Χάνς Πίτερ Μάιερ συμφώνησε, μια που είναι πιο παλιός ε, εδώ, να αναλάβει την Προεδρία για να μπορέσω εγώ να πάω και να συναντηθώ με την κυρία Ρέντινγκ. Θα φροντίσουμε να γίνει η αλλαγή αυτή όπως πρέπει. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Έρχομαι τώρα λοιπόν στο πρόγραμμα δράσης για τα τελωνία. Έχει να κάνει με την διάκριση που κόβουμε σε δύο μέρη δηλαδή το φίσκους. Ο κύριος Μπαλτασάρη είναι ο εισηγητής μας. Θα δούμε τις τροπολογίες, τις συμβαστικές τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Ο κύριος Καπαράτη είναι από τους σοσιαλιστές, Σμίτ από τους φιλελεύθερους, δεν ξέρω, δεν βλέπω εδώ πέρα άλλους και όδες εισηγητές. Οπότε ο κύριος Βαλταζάρη παρακαλώ να μας ενημερώσει, να μας μιλήσει και για τους συμβιβασμούς που προτείνονται και μετά θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές και θα δούμε μετά τι θα κάνουμε. Ο κύριος Δασκάλου είναι εδώ, που είναι επικεφαλής τμήματάρχης και εκείνο παρακαλώ να σχολιάσει. Ο κύριος Βαλτασάρη τώρα εισηγητής, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος υπό την έννοια ότι μετά από την ανάλυση των 40 τροπολογιών που υποβλήθηκαν στο σχέδιο έκθεσης, αποφάσισα να καταλήξω και να επεξεργαστώ τρεις συμβιβαστικές τροπολογίες. Υπάρχουν άλλοι, άλλοι, άλλες 20 τροπολογίες και οι υπόλοιπε θα ψηφιστούν όλες μαζί. Η θέση μου είναι υπέρ όλων των τροπολογιών, εκτός όπως ήδη το είπα στην προηγούμενη συνεδρίασή μας, είναι της κυρίας Πατρίτσια Μπάρντε Κάμεν, που έχει να κάνει με τις υποψήφιες χώρες, ε, τις πιθανές υποψήφιες χώρες και τις χώρες που είναι στη διαδικασία της ένταξης. Ε, υπάρχει ο γενικός στόχος του προγράμματος, άρθρο 6, Υπάρχει το άρθρο για, τις, ε, για τους γενικούς σκοπούς του προγράμματος, το άρθρο 6 για τους ειδικού σκοπούς του προγράμματος και το άρθρο για τον ε, τελικό σκοπό του προγράμματος. Δεν υπήρχαν ιδιαίτερες ε, διαφορές, ασυμφωνίες ως προς την επαναδιατύπωση της νέας έκθεσης για την κυρία φορολογία. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν δυσκολίες. Αυτό προβλέπω. Βρίσκομαι εδώ ε, να ακούσω τα τυχόν τελευταία σχόλια από τους σκιώδεις εισηγητές και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ όλους για τη συμβολή σας, για τις προτάσεις, τις υποδείξεις που εμπλούτησαν αυτήν την έκθεση. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοφεράτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Μπαλτάσαρε για την ε, εξαιρετική δουλειά του, για τους συμβιβασμούς που μας πρότεινε, για τις λύσεις που μας βρίσκουν σύμφωνους. Όπως είπε και ο ίδιος επί της ουσίας, ε, ε, αλλά και λόγω της καλής μας συνεργασίας, έχουμε καταλήξει σε μία ομόφωνη και απλή λύση. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα της δουλειάς μας θα τύχει ομοφωνίας και θα μας βοηθήσει στο μέλλον, ιδίως αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να ακούσει τις προτάσεις μας ε, για την ανάπτυξη των τεχνικών ικανοτήτων, τη χρήση της πληροφορικής. Επίσης για το μέλλον σημαντική θα είναι η πρόθεση της συγκριτικής ανάλυσης των τελωνίων με, με τρόπο ο οποίος θα είναι αξιόλογος. Θέλω να τονίσω ότι οι πόροι ε, αυτού του προγράμματος στο τέλο της συζήτησης για τους πολιετής δημοσιονομικούς πόρους έχουν αυξηθεί. Θετικό το αποτέλεσμα. Καλό είναι να μην βρεθούμε μπροστά σε ανεπάρκεια πόρων. Φυσικά αυτό δεν εξαρτάται από μας, αλλά επειδή έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά, θα πρέπει να έχουμε και τα μέσα να την υλοποιήσουμε στην πράξη. Θα πρέπει να έχουμε τους αντίστοιχους πόρους. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ραφαέλε καθώς και τους άλλους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Μπαλτασάρε, τον εισηγητή. Ξέρουμε όλοι ότι παρόλο που δεν είναι το θέμα το πιο σεξι στην ημερήσια διάταξη, είναι βεβαίως πάρα πολύ σημαντικό, κυρίως στις μέρες μας όπου χρειαζόμαστε όλα τα έσοδα τα οποία μπορούμε να έχουμε. Και χαίρομαι που μπορώ να πω ότι έχουμε καταλήξει σε πολύ καλούς συμβιβασμούς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Το μόνο πράγμα και αυτό είναι ίσως κάτι όπου θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό η συμφωνία γι' αυτό είναι ότι δεν θα έπρεπε να περιλάβουμε στην χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξοπλισμούς όπως σαρωτές ή όργανα εργαστηρίου. Μπορούμε να βρούμε αλλού πόρους χρηματικούς για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο να μπορούν όλοι να συμμετάσχουν στα συστήματα, τα μηχανογραφικά, στην τεχνολογία πληροφορικής που να λειτουργεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτό είναι το ουσιαστικότερο πράγμα το οποίο θα πρέπει να επιτύχουμε στο μέλλον. Αυτή, αυτή είναι η μόνη παρατήρηση που έχω να κάνω. Έχω κάποιες επιφυλάξεις ως προς τη χρηματοδότηση άλλων μέσων, εκτός που δεν ανήκουν στον τομέα των πληροφοριών των επικοινωνιών. Ευχαριστώ. Ε, μήπως θέλει κανένα άλλο μέλος ε, να λάβει το λόγο πρωτού δώσω το λόγο στην Κομισιόν για να μας δώσει τις απόψεις της σχετικά με το πρόγραμμα αυτό. Πολύ καλά. Ο κύριος Δασκάλου έχει το λόγο, θα μπορούσε να μας πει την άποψή του. Σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μπαλτασάρη και το σκιώδη συγητή για αυτήν την εκδοχή. Την έλαβα πολύ αργά και δεν είχα το χρόνο να διαβάσω όλο το κείμενο. Θα σας πω απλώς μερικά πράγματα για το τι συνέβη στο Συμβούλιο. Είχαμε μια συμφωνία στο Συμβούλιο ε, με την εκδοχή το σχέδιο κανονισμού που μπορεί να υιοθετηθεί με πάρα πολύ μικρές αλλαγές, τεχνικές αλλαγές. Οι στόχοι και οι γενικές αρχές παραμένουν ως προτάθηκαν από την Επιτροπή και αυτό που είναι σημαντικό για την Επιτροπή αυτή είναι να ξέρει ότι αρχικά ορισμένα κράτη-μέλη ζήτησαν το πρόγραμμα να χρηματοδοτεί και τον εξοπλισμό και μετά από συζήτηση αποφασίστηκε να εγκατελειφθεί αυτή η ιδέα, αυτό το αίτημα και παρά να έχουμε πρόνοιες για την χρηματοδότηση του εξοπλισμού, εισήγαγαν ε, μια δήλωση ε, στα πρακτικά του Συμβουλίου με σύσταση στην Κομισιό να κάνει μια μελέτη ούτως ώστε να προσδιοριστούν μέσα για την χρηματοδότηση του εξοπλισμού για την επόμενη γενεά του πολιετούς δημοσιονομικού ε, πλαισίου και θα είναι έτοιμο αυτό το 2018. Αυτή είναι η κατάσταση που αντιστοιχεί με την θέση της Κομισιόν σχετικά με τον εξοπλισμό, δηλαδή ότι ο εξοπλισμός θα πρέπει να χρηματοδοτείται από άλλα προγράμματα ε, και όχι από το πρόγραμμα Τελωνία 2020 και είναι από τα βασικά σχόλια τα οποία είχαμε και αναφέραμε επίση και στην προηγούμενη συνεδρίαση. Αυτά είναι όσα είχα να πω κύριε Πρόεδρε. Πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπαλτασάρε, έχετε άλλα σχόλια να κάνετε σχετικά με το θέμα αυτό. Έχουμε τι ε, τις, τις τροπολογίες συμβιβασμού. Οι τριπολογίες συμβιβασμού έχουν, α, ε, έχουν ε, δημοσιευθεί μαζί με την κατάλογο ψηφοφορίας. Θα σας ζητήσω ίσως να διανεμηθούν αυτές. Έχετε σχόλια να προσθέσετε κύριε Μπαλτασάρε, απαντώντας στην Κομισιόν και στους συναδέλφους σας, για να μας προσανατολίσετε προς την ψηφοφορία που θα λάβει η χώρα αύριο το απόγευμα. Ναι. Πιστεύω ότι κατ' ουσίαν δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Ευχαριστώ πολύ για τις απόψεις και για τα θετικά σχόλια. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτή την τελευταία πτυχή που αφορά τη χρηματοδότηση και τις υποδομές. Αλλά κατά τα λοιπά, όλα τα λοιπά μας βρίσκουν σύμφωνους και δεν υπάρχουν περαιτέρω σχόλια από την πλευρά μου. Ευχαριστώ. Good. Okay, well... Ωραία. Έτσι ε, θα κλείσουμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενο θέμα, αλλά η κυρία Λεγκρίπ, η συγγήτρια, δεν είναι εδώ. Ε, ούτε και εκπρόσωπος της Επιτροπής σχετικά. Μάλιστα. Επομένως, σας κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για τσάι μέχρι τις 4 και 4. Εκτός κύριε Σουβάπαν, θα θέλατε να πείτε κάτι... Α, κύριε Κοφεράτη ε, αναρωτιόμουν αν θα μπορούσαμε να περάσουμε απευθείας στην έκθεση του κυρίου Σβάμπ. Γιατί όχι, γιατί να μην συζητήσουμε απευθείας την έκθεση του κυρίου Σβάμπ. Έρχεται η κυρία Λεγκρίπ, της μιλήσατε. Εντάξει, θα τη τηλεφωνήσουμε. Και, ε, μας λένε ότι και από την Επιτροπή είναι καθοδόν. Οπότε και πάλι προτείνω να πιούμε ένα φλιτζάνι τσάι και να περιμένουμε μέχρι να φτάσει η κυρία Λεγκρίπ. liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, lassen Sie uns fortfahren. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε μετά από αυτή την μικρή διακοπή. Περνάμε στο επόμενο σημείο, που είναι το σημείο 4, για την αναδιατύπωση του ενωσιακού τελωνιακού κώδικα. Η συγκήτριά μας είναι η κυρία Κωνστάνσο Λεγκρίπ που ήρθε, οπότε θα τη δώσω το λόγο ευθύ αμέσω. Παρακαλώ, κυρία Λεγκρίπ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα είμαστε εδώ για να εξετάσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες που υπέβαλα στους σκιώδεις εισηγητές και τις οποίες θα συζητήσουμε σήμερα για την αναδιατύπωση του Ενωσιακού Τελωνιακού Κώδικα. Μετά από εβδομάδες ε, Συζητήσουν μεταξύ μας, ανταλλαγών μεταξύ μας για μια τόσο περίπλοκη και δύσκολη υπόθεση, έχουμε καταλήξει κάπου και είναι περίπλοκη γιατί έχει να κάνει βλέπετε με την καθημερινότητα των τελωνίων μας και με την καθημερινότητα των οικονομικών φορέων μας, των εγκεκριμένων ε, κλπ. Επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, το πώς δηλαδή θα βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των τελωνίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι κάτι πολύ βασικό για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, βασιζόμαστε στον ε, ε, τελωνιακό κώδικα του 1992. Εννοείται ότι έκτοτε υπάρχουν πολλές νομοθετικές πράξεις που έχουν υιοθετηθεί, έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα, οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά πρότεινε πριν από λίγους μήνες να αντικαταστήσουμε τον κανονισμό 450 του 2008, που τον λέμε εξεχωρισμένο το λιωνιακό κώδικα από έναν άλλον αναδιατυπωμένο, ο οποίος να ανταποκρίνεται στους στόχους που μας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο που μας πέρασε και τους επιθυμίζω τους στόχους αυτούς. Πρώτον, να αναβληθεί η ημερομηνία εφαρμογή όσον αφορά τον τολυνικό κώδικα. Δεύτερον, να προσαρμοστεί η βάση της ε, θέσης ισχύ της εθήκη τη Λισαβόνας και τρίτον, να λυθεί υπόψη όλες οι ρυθμίσεις του Τελωνιακού κώδικα που έχουν να κάνουν με τον εξυγχρονιασμό τη πληροφορικής, με την ασφάλεια κλπ. Θα σας πω τώρα και δύο λόγια για το πώς έχουν προχωρήσει οι εργασίες από πλευράς του Συμβουλίου. Πιστεύουμε ότι η εμβάθυνση του τελωνιακού κώδικα είναι κάτι που πρέπει να συνεχιστεί είναι, πρόκειται για ένα κοινοτικό κεκτημένο πολύ βασικό. Οι υπουργοί λοιπόν που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ανταγωνισμού στις 11 Δεκεμβρίου πριν από λίγες μέρες δηλαδή συνεδρίασαν και επανέλαβαν την βούλησή τους για έγκριση της ε, συμφωνίας αυτής για αναδιατύπωση του τολωνιακού κώδικα πριν από τον Ιούνιο του 2013. Και είναι καλό που επανέλαβαν τη βούλησή τους σε αυτή στο Συμβούλιο. Η Ιρλανδική Προεδρία τώρα που θα αναλάβει και θα πάρει τη σκητάλη από την Κυπριακή Προεδρία τον Ιανουάριο. Η Ιρλανδική Προεδρία λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό για να προχωρήσει το θέμα αυτό και έτσι μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου του 2013 να έχουμε μια κοινή πρόταση που θα μας υποβάλει το Συμβούλιο. Και θα μπορούμε έτσι να λάβουμε υπόψη μας τις προθεσμίες. Πάντως όσον αφορά εμάς Κοινοβούλιο κάναμε τα πάντα για να προχωρήσουμε με καλό ρυθμό. Και έτσι πιστεύω ότι μπορούμε να προβλέψουμε την άνοιξη που μας έρχεται να εγκρίνουμε στην Ολομέλεια το νέο αυτό τελωνιακό κώδικα, την αδιατύπωση δηλαδή. Τώρα όλο αυτό τον καιρό, γιατί εγώ σας παρουσίασα την έκθεσή μου αμέσως μόλις γυρίσαμε από τις καλοκαιρινές διακοπές το Σεπτέμβριο. Ε, λοιπόν, κάθε φορά θέλησα να συμμετέχουν εκεί οι σκιώδεις εισηγητές από όλες τις πολιτικές ομάδες για να καταλήξουμε σε μια πολιτική γραμμή που να είναι κοινή και σαφής. Το πολιτικό μήνυμα λοιπόν, το κοινό μεταξύ μας, σκιωδών εισηγητών δηλαδή και εμού της ίδιας, είχε ως εξής. Πρώτον, απλοποίηση και διευκόλυνση για τους οικονομικούς φορείς, ξεκινώντας βέβαια από τους συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς που είναι πολύ άριθμοι, όλο και περισσότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν ένα οικονομικό πλαίσιο, όπως καταλαβαίνετε, αρκετά δύσκολο αυτή την εποχή. Ασφάλεια λοιπόν και διευκόλυνση απέναντι σε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Σιγουρία και ασφάλεια λοιπόν. Έπειτα εξυγχρονισμός της υπάρχουσας νομοθεσίας, εννοείται. Αλλά επίσης, και αυτό είναι ένα νέο πολιτικό μήνυμα δικό μας, σεβασμό των προνομίων και των αρμοδιοτήτων των διαφόρων ευρωπαϊκών θεσμών. Έχω την αίσθηση ότι καταφέραμε και δουλέψαμε με διαφάνεια και επικοδομητικά. Και γι' αυτό θέλω θερμά να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδες εισηγητές που βοήθησαν τόσο πολύ για το θετικό τους πνεύμα, για τη συνεργασία τους, προκειμένου να καταλήξουμε εδώ που καταλήξαμε. Αυτή η καλή θέλησή τους και η πικοδομητική δουλειά που κάνανε, με διαφάνεια πάντα, είναι και αυτό το οποίο μας καθοδήγησε και τις τελευταίες εβδομάδες και με βοήθησε και εμένα να καταλήξω στις συμβαστικές τροπολογίες που σας έχω υποβάλει και τις οποίες θα σας παρουσιάσω κάπως σύντομα. Δεν είναι πάρα Υπάρχουν διάφορες τροπολογίες λοιπόν για θέματα πολύ σημαντικά. Θα σας παρουσιάσω τις δύο συμβιβαστικές λοιπόν που θέλω και να σας υποβάλω. Η πρώτη έχει να κάνει με το άρθρο 62 παράγραφος 4 και ορίζει την αξία στο τελωνείο. Η συμβαστική τροπολογία που σας υποβάλλω εγώ σήμερα, που είναι η α, συμβαστική μου α, έχει ως στόχο να συμβιβάσει κατά κάποιο τρόπο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο της τροπολογίας που είχαν υποβληθεί νωρίτερα από δύο συναδέρφους μας, η 84 δηλαδή του κυρίου Σουβάμπ, και η 97 του κυρίου Σμιτ. Είναι δύο τροπολογίες αυτές που προσπάθησα να παντρέψω. Ε, προσφέρουν διευκρινήσεις, είναι συμπληρωματικές για τον τρόπο με τον οποίο η τελωνιακή αξία καθορίζεται. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν κατέληξα και εγώ στην συμβαστική μου τροπολογία λαμβάνοντας υπόψη μου ότι πρόκειται για συμπληρωματικές τροπολογίες. Η συμβαστική μου λοιπόν α μιλάει για τον καθορισμό της τελωνική αξίας, αξία στο τελωνίο, βάσει ενό συγκεκριμένου ορισμού και ισορροπημένου. Η δεύτερη συμβαστική τροπολογία μου, η β, έχει να κάνει με το άρθρο 181 παράγραφος 3 σημείο 2 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το άρθρο λοιπόν αυτό 181 αναφέρεται στις προϋποθέσεις για τους συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς. Και αυτή η συμβαστική τροπολογία Β συγκεντρώνει σε μία μόνο τροπολογία τρεις προηγούμενες τροπολογίες που έχουν υποβάλει συνάδελφοι ή 32 που εξάλλου εγώ ίδια είχα διατυπώσει αλλά και την 172 και την 171, 162 και 171 του κ. Σμιτ. Είναι η συμβαστική μου αυτή τροπολογία, λοιπόν, έχει σαν στόχο την, ε, την αξιοποίηση του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα. Για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία η αναγνώριση και η αξιοποίηση του καθεστώτος αυτού του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα ευχαρίστως να ακούσω ότι έχουν να πούν οι σκιώδεις εισηγητές και τι παρατηρήσεις έχουν να κάνουν πάνω στις συμβαστικές μου τροπολογίες. Κατάλαβα ότι ίσως να υπάρξει από κάποιον μια ελαφρά επιφύλαξη από μια πολιτική ομάδα για κάποιες ε, λέξεις που περιλαμβάνει η τροπολογία μου, η συμβαστική Β. Πάντω, στόχο τη συμβαστική αυτή τροπολογία Β είναι να αξιοποιήσει το καθεστώ του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι ένα θεμελιώδες ε, μήνυμα για τις επιχειρήσεις μας, τις μικρές και μεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες πολύ συχνά και το έχουμε δει, γιατί όλοι μας ήρθαμε σε επαφή με οικονομικούς ε, φορείς εγκεκριμένους, έχουν την αίσθηση μερικές φορές ότι δεν έχουν ιδιαίτερα ωφέλη από το καθεστώς αυτό εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, παρά τη δουλειά που έχουν, να κάνουν, που έχουν να κάνει μέχρι τώρα για να πετύχουν αυτό το καθεστώς του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα. Οπότε, όλες οι πολιτικές ομάδες πρέπει να δείξουν την ε, καλή τους θέληση για να αξιοποιηθεί όσο γίνεται περισσότερο το καθεστώς ε, αυτό από τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς. Πρέπει να αποτελεί την είσοδο σε μια διευκόλυνση που τους προσφέρουμε όσον αφορά την είσοδο στα τελωνία. Τώρα υπάρχουν και δύο προφορικές τροπολογίες που υποβάλλω για να τις αξιολογήσετε και να τις εγκρίνετε. Μία πρώτη μικρή προφορική τροπολογία θέλει να διαγραφεί παράγραφος H στην τροπολογία μου 14, του σχεδίου δηλαδή έκθεσής μου, επειδή, πώς να σας το πω, θέλαμε εδώ να έχουμε κάποια συνοχή κατά προτίμηση. Η τροπολογία 14, πρέπει να ξέρετε, στην παράγραφο Age, ε, δίνει την αρμοδιότητα για κατεξοδότηση πράξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να ε, μπορούν εύκολα να υποφεληθούν οι εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς, αλλά εγώ Θέλω να διαγραφούν όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στη δυνατότητα άρσης της υποχρέωσης, εγκατάστασης στην επικράτεια για τους συγκεκριμένου ε, αυτούς οικονομικούς φορείς, έπρεπε να γίνει μια μικρή διόρθωση. Αυτή είναι η πρώτη μικρή προφορική τροπολογία. Να βγάλουμε δηλαδή τη μικρή παράγραφο H. Στη δεύτερη προφορική μου τροπολογία έχει να κάνει με το 164 παράγραφος 3 του κανονισμού. Αυτή η δεύτερη προφορική τροπολογία λοιπόν έχει ως στόχο να διευκρινίσουμε ποια στιγμή ε, αποδεχόμαστε τη γραπτή δήλωση του εισαγωγέα προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη απλοποίηση γιατί αυτό είναι πάντα ο στόχος. Και θα ολοκληρώσω με το λεπτό θέμα των εκτελεστικών πράξεων και των κατεξουσιοδότηση πράξεων, που είναι ευαίσθητο, το ξέρω. Από την αρχή που ασχολούμαι με το θέμα αυτό, καταλαβαίνω ότι αυτό το θέμα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και η κατανομή αρμοδιοτήτων ε, ανάμεσα στα θεσμικά όργανα που απορρέουν από το άρθρο 190 και 191 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ συχνά με τους σκιώδεις εισηγητές το συζητήσαμε αυτό το θέμα. Και πιστεύω ότι είναι ζωτική σημασία να έχουμε μια θέση με συνοχή και να στηρίξουμε τη θέση μας, την οποία πιστεύω ότι τη συμμεριζόμαστε όλοι εδώ σε αυτήν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Και ποια είναι αυτή η θέση μας είναι η προώθηση των αρμοδιοτήτων και των προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή είναι και η θέση που εκφράζω εγώ επανειλημμένως στο σχέδιο εκθεσής μου και θα το βρείτε και στις τροπολογίες των συναδέλφων. Κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου το επαναλαμβάνουμε. Θα το επαναλάβουμε ξανά και ξανά. Θα αρχίσει μάλλον τέλη Ιανουαρίου. Θέλουμε οι συζητήσεις να είναι ζωντανές και για αυτό το θέμα, το τόσο λεπτό και ευαίσθητο των αρμοδιοτήτων πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό ο καθένας μας να κάνει τις προσπάθειες φυσικά που χρειάζεται και επιβάλλεται, αλλά με κάποια ισορροπία και με σεβασμό στις συνθήκες και στις αρμοδιότητες έτσι όπως αυτές αναγνωρίζονται για το κάθε θεσμικό όργανο. Έτσι θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί πιστεύω γιατί έτσι θα πετύχουμε περισσότερη οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα για τις ευρωπαϊκές μας επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Äh, äh, ευχαριστώ πολύ. Είναι αλήθεια ότι είναι ένα θέμα αρκετά περιπλοκό και βλέπουμε ότι ασχολήθηκες διεξοδικά με όλα τα θέματα αυτά. Και στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας είναι σημαντικό να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στις κατεξουσιοδότηση πράξεις και τις εκτελεστικές πράξεις, διότι έχουμε στο επίπεδο αυτό μια ευθύνη και αρμοδιότητα και πρέπει να δούμε τι εξαρτάται από τη δική μας αρμοδιότητα. Πρωτού δώσω το λόγο στο σκιώδη συγητή, θα ήθελα να καλωσορίσω μια ομάδα επισκεπτών που έρχονται από την δική μου περιφέρεια, 12 εκπαιδευτικοί, από ένα σχολείο και είμαι πάρα πολύ ευτυχής που βλέπω ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί άντρες και γυναίκες που ασχολούνται με τα όσα συμβαίνουν εδώ για να τα διδάξουν μετά στα, ε, στους μαθητές τους. Και τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην Σιλβάνα Ράπτη. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ επίσης και την εισηγήτρια, την κυρία Λεγκρίπ. Ξέρετε, κάθε φορά στις εκθέσεις εδώ όταν συζητάμε αρχίζουμε τις ευχαριστίες. Ε, θέλω να υπογραμμίσω ότι νιώθω απόλυτα την ανάγκη να πω ένα γνήσιο, πραγματικό, αληθινό ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Και το υπογραμμίζω γιατί ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε μέσα στο Κοινοβούλιο θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικός και γιατί μας βοηθάει να καταλήξουμε στα καλύτερα δυνατά συμπεράσματα για τους ευρωπαίους πολίτες για τους οποίους εργαζόμαστε αλλά και γιατί ταυτοχρόνως δίνουμε ένα παράδειγμα αν μπορώ να το πω έτσι για το πώς μπορούμε να εργαζόμαστε για μια καλύτερη Ευρώπη. Έτσι λοιπόν δεν έχω να πω πολλά, έχω να πω ελάχιστα και αυτό με χαροποιεί έτσι ε, έχω να ε, επιμείνω λιγάκι στο θέμα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα. Το είπε πάρα πολύ ωραία η κυρία Λεγκρίπα ότι ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ακριβώς γι' αυτό θέλουμε τον εγκεκριμένο οικονομικό φορέα να τον διευκολύνουμε. Ακριβώς όμως επειδή οι διευκολύνσεις που δίνουμε είναι πολύ σοβαρές, είναι πολύ σημαντικές. Θέλουμε ταυτοχρόνως να έχουμε και εμπιστοσύνη σε αυτόν τον οποιονδήποτε εγκεκριμένο οικονομικό φορέα. Τα λέω όλα αυτά για να καταλήξω ότι ε, τα κριτήρια με βάση τα οποία κάποιος αποκτά το καθεστώς του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα πρέπει για μας να είναι στο σώμα του κώδικα. Ε, έτσι λοιπόν έχω μία, πώς να το πω, δεν, δεν, ε, δεν, μπορώ λιγάκι να καταλάβω γιατί η αναθεώρηση των κριτηρίων θα πρέπει να εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, την καταθέτω τη σκέψη αυτή. Ασφαλώς είμαστε σύμμαχοι με την Επιτροπή, η οποία ρυθμίζει πολλά άλλα θέματα για τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς και το καταλαβαίνουμε απολύτως. Αλλά τα κριτήρια και η αναθεώρησή τους θα πρέπει να ρυθμίζονται σαφώς. Ε, σε αυτό το σημείο θα υποβάλουμε μία προφορική τροπολογία. Και καταλήγω ε, με μία ακόμη ευχαριστία, όπως ξεκίνησα. Ευχαριστώ την εισηγήτρια που έχει δεχτεί την άρση της δυνατότητας να είναι η εγκεκριμένη οικονομική φορείς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βάζω μια τελεία, ευχαριστώ και πάλι και νομίζω ότι και στη συνέχεια η δουλειά μας θα είναι ε, το ίδιο καρποφόρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στον ε, Όλο Σμίτ, εκπρόσωπο των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λεγκρίπ, την εισηγήτρια, η οποία υπήρξε πάρα πολύ φιλόδοξη και έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ε, με όλη της την καρδιά και ελπίζω να μπορέσουμε να κατακαλύξουμε ε, σε δίκαιο συμβιβασμό. Δεν είναι πρόβλημα για μένα να υποστηρίξω ένα συμβιβασμό και πιστεύω ότι υπάρχουν ισορροπημένοι συμβιβασμοί. Το μόνο πράγμα το οποίο με κάνει να αμφιβάλλω λίγο είναι η πρόταση να διαγράψουμε την προσωρινή εναπόθεση και πρόκειται για το άρθρο 101.3.4. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι επωφελές για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και πιστεύω ότι αυτό απαιτεί πολύ ερμηνεία για να ξέρει κανείς ποια διασάφηση θα υποβάλει. Ε, αμφιβάλλω, δεν ξέρω βεβαίως αν ε, έχω δίκιο, αν είναι ο καλύτερος τρόπος αυτός. Και τελευταίο πράγμα, διότι και εγώ θέλω να είμαι πολύ σύντομος, πιστεύω ότι οι κανόνες της μη προτιμησιακής καταγωγής δεν έχουν μεγάλη σημασία για τα τελωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχω, δεν ξέρω, έχω κάποιες υποψίες, καχυποψίες και αμφιβολίες. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι μια κρυμμένη ατζέντα, μια συγκαλυμμένη ατζέντα διότι αυτή η πρόταση, αυτή η νομοθετική πρόταση θα πρέπει να είναι σαφής, να έχει σαφείς κανόνες και ορισμούς. Αυτή είναι μια έκκληση κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Λογκρίπ επίσης. Ναι, για τους πράσινους και εγώ θα είμαι πάρα πολύ ε, σύντομη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και οφείλω να ομιλογήσω ότι πρέπει να είμαι ειλικρινής και έντιμη μαζί σας διότι είδαμε ότι υπήρχαν μεγάλες διχογνωμίες από τα λόμπι, υπάρχουν διάφορα συμφέροντα που αντιπροσωπεύονται και πρέπει να σας ευχαριστήσω διότι πετύχατε ένα καλό ισορροπημένο συμβιβασμό και θα πρέπει όλοι να μπορούν να δεχθούν το κείμενο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι αυτό ήταν το έργο το σημαντικότερο για έναν εισηγητή να καταλήξει σε μια ισορροπία την ε, πετύχατε αυτήν την ισορροπία. Υποστηρίζουμε ε, τις τροπολογίες αυτές, τους συμβιβασμούς αυτούς ε, και είπα ότι συμφωνούμε με τις νέες συμβιβαστικέ τροπολογίες σας και συμφωνώ με τον κύριο Σμιτ. Πιστεύω ότι θα πρέπει επίσης να δούμε πώς τα πράγματα λειτουργούν σε αυτό το επίπεδο και να δούμε τι γίνεται με αυτήν την μη προτιμησιακή καταγωγή διότι είναι ένα ευαίσθητο λεπτό θέμα και υπάρχουν ορισμένα στοιχεία συγκαλυμμένα τα οποία θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπίλαν για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Λεγκρίπα για την τέλεια εργασία της για τον τέλειο τρόπο που εργάστηκε πάνω σε αυτή την έκθεση και θα είμαι σύντομος γιατί υπάρχει συμφωνία ως προς τα περισσότερα θέματα σύμφωνα με τις συζητήσεις που έγιναν με τους σκιώδεις εισηγητές. Δύο συμβιβαστικές τροπολογίες, τροπολογία 8 για την τελωνιακή αξία, για τον τρόπο καθορισμού της τελωνιακής αξίας και τροπολογία Β, <clears throat> άρθρο 181 υπό παράγραφος 3. Όσο αφορά την τροπολογία 1, πιστεύω ότι θα αφορά σωστά την προτιμησιακή μεταχείριση και η ομάδα μου θα την υπερψηφίσει. Για την τροπολογία Β θεωρούμε ότι είναι μια καλή πρόταση. Ωστόσο, εμείς έχουμε προτείνει να απαλληφθούν οι τελευταίες λέξεις, δεν απαιτούνται περαιτέρω έλογχοι, γιατί η διατύπωση αυτή μπορεί να δημιουργήσει ανώφελα προβλήματα ερμηνείας του άρθρου αυτού και θα ήταν κρίμα. Θα ήταν κρίμα να μην γίνει δεκτή αυτή η πρότασή μας. Για το λόγο αυτό δεν μπορούμε να στηρίξουμε τη συγκεκριμένη συμβιβαστική τροπολογία και θα απόσχουμε κατά την ψηφοφορία. Γενικά όμως θα στηρίξουμε την 171 του κυρίου Σμιτ που πιστεύουμε ότι είναι η πιο σαφής και όσο αφορά την προφορική υπαριθμών 2 θα στείλω την ελαφρώς τροποποιημένη πρότασή μου στην εισηγήτρια και θα αναμείνω τα σχόλιά της. Ελπίζω ότι η πρότασή μας θα γίνει δεκτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και τη συμβολή σας. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ε, για την εκ μέρους της Γκουε υπάρχει κάποιος όχι. Έλαβα μία, ένα αίτημα για τους φιλελεύθερους δημοκράτες, αλλά δεν βλέπω κανέναν στην αίθουσα. Στη συνέχεια δίνω τον λόγο στον κύριο Τσιρίνσκι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν θέλω να επαναλάβω όσα υπόθηκαν, αλλά θα ήθελα και εγώ να πω ευχαριστώ πάρα πολύ στην κυρία Λεγκρίπ, καθώς και στους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, ήταν πολύ πετυχημένη η εργασία αυτή. Δεν μπορώ να πω ότι συμφωνούμε με όλα. Ε, γιατί χρειάζομαι την άδεια του Προέδρου του Σώματος για να το πω αυτό, αλλά πάντως ακολουθούμε την ίδια γραμμή σκέψης. Ίσως όχι στα πάντα. Ε, υπάρχουν και κάποιες λεπτομέρειες που θα ξεκαθαριστούν στον τριμερή διάλογο. Ε, δεν, όπως σας είπα, δεν είμαι εξουσιοδοτημένος να σας πω ότι συμφωνούμε, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι υιοθετούμε τον ίδιο τρόπο σκέψης. Θα παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας και στις άλλες υπηρεσίες και στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα κλείσω λοιπόν την παρέμβασή μου και θα σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κανείς εκ μέρους του Συμβουλίου να πάρει το λόγο, επομένως δώνω εκ νέου των λόγων στην κυρία Λεγκρίπ, την εισηγήτρια, για να κλείσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα για άλλη μια φορά πραγματικά και ειλικρινά να εκφράσω τις ε, θερμές ευχαριστίες μου, τις θερμότατες ευχαριστίες μου στους σκιώδεις εισηγητές, οι οποίοι με βοήθησαν πάρα πολύ με τις προτάσεις τους, με τη δουλειά τους, ε, με την ενθάρρυνσή τους, με τα κίνητρα και την κινητοποίησή τους. Ε, και έτσι πραγματικά ε, εποφελήθηκα από όλα, από τις υποδείξεις τους, ε, από τα σχόλιά τους. Ε, παρέλειψα να αναφέρω, σφάλμα δικό μου, να αναφέρω το θέμα των κανόνων για την προέλευση. Ένα πολύ ουσιώδες θέμα. Ε, είναι σημαντικό ε, ο ορισμός που θα δώσουμε να υπάρξει στο βασικό κείμενο, να είναι μέρος του βασικού κειμένου. Υπάρχουν πολλές εκδοχές, είναι αλήθεια, έχουν προταθεί πολλές εκδοχές. Εγώ προτείνω μια έναν συγκεκριμένο ορισμό στην τροπολογία 19 του σχεδίου έκθεσης. Πρόκειται για έναν ορισμό για τους κανόνες προέλευσης για τον κανόνα προέλευσης που προέρχεται από τη Συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Θεωρώ ότι έτσι υπάρχει κάποια νομιμοποίηση για την υιοθέτηση του ορισμού αυτού. Αναγνωρίζω όμως ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, ε, θεμητές ε, οι οποίες θα συζητηθούν όλες. Να πω όμως ότι στη δική μου απόπειρα προσπάθησα να δώσω τον ορισμό που είναι πιο κοντά στα ισχύοντα νομοθετικά κείμενα που την χάνουν διεθνούς αναγνώρισης. Θεώρησα ότι αυτός είναι ο πιο σωστός τρόπος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και έτσι ολοκληρώνουμε και το σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Το επόμενο σημείο εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων έχει αναβληθεί. Η συζήτηση για το θέμα αυτό έχει αναβληθεί. Επομένως, σημείο 6 θα το, θα το συζητήσουμε επρόκειτο να το συζητήσουμε αργότερα, αλλά εφόσον είναι εδώ ο εισηγητής, ας το συζητήσουμε. Δίνω το λόγο στον κύριο Σβάμπ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα θέλω να διευκρινίσω ότι οι παρεμβάσει των συναδέρφων έτσι κι έχουν βοηθήσει πολύ να βελτιωθεί το κείμενο. Και μια που πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα, α είμαστε ειλικρινεί. Δεν είναι εύκολο πάντα να ε, επανακαλύψουμε την ε, τον τροχό όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών στην Ευρώπη και την πολιτική ανταγωνισμού. Επικεντρωθήκαμε λοιπόν σε κάποια βασικά στοιχεία και νομίζω τα καταφέραμε. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα το εξή. Με ποιο τρόπο μπορούμε να κρίνουμε τη συγχώνευση δύο μεγάλων επιχειρήσεων στον τομέα των ε, αποστολών Express, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Υπάρχουν συνάδελφοι εδώ οι οποίοι δεν επιθυμούν να αναφερόμαστε σε επιχειρήσεις ανταγωνιστικές. Ε, μπορώ να το καταλάβω και γι' αυτό και μπορούμε να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάποιο συμβιβασμό. Ας πούμε το ότι πήρε την TNT UPS μπορούμε να το αναφέρουμε χωρίς να αναφέρουμε τα ονόματα. Δηλαδή να πούμε ότι είναι αναγκαίο οι διατλαντικές συγχωνεύσεις να επιτρέπονται, αλλά υπό αντίστοιχες προϋποθέσεις. Επίσης ότι πρέπει κάποιος ρυθμιστής να καλύπτει και τις δύο επιχειρήσεις, κάτι το οποίο δεν ισχύει σήμερα. Μεγάλες ευρωπαϊκές ή γερμανικές επιχειρήσεις είναι παρούσες στην Αμερικανική αγορά, αλλά αναγκάστηκαν να παραχωρήσουν αγορές και άλλες επιχειρήσεις που θέλησαν να εγκατασταθούν στην Ευρώπη υπάρχουν. Το θέμα δεν είναι να κλειστεί η Ευρώπη και να υπερπροστατεύεται, όχι, πρέπει να είναι ανοιχτή βέβαια στον υπόλοιπο κόσμο, όταν όμως μεγάλες επιχειρήσεις θέλουν να εγκατασταθούν και γίνεται κάποια συγχώνευση, πρέπει να έχουν την δυνατότητα να έχουν το κομμάτι της ε, αγοράς που τους πρέπει, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεγάλες ε, παγκόσμιες δυνάμεις. Τέλο πάντων, καταλήξαμε και με τον κύριο Χάρμπορ σε κάποια συμβιβασμό. Και έχουμε και την τροπολογία του κύριου Οντί. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω καταλάβει πάρα πολύ καλά την τροπολογία του και γι' αυτό ακριβώς και είπα ότι δεν μπορώ να συστήσω την έγκριση της τροπολογίας αυτής και ότι θα πρέπει να την συζητήσουμε. Ο κύριος Κοφεράτη τώρα από τη δικιά του την ε, πλευρά, όπως και για την ε, διαχείριση της εσωτερικής αγοράς, σύντομα θα σας πω, ότι ήταν διατεθειμένος για συμβιβασμό. Και τι λέει τελικά, λέει ότι θέλουμε να έχουμε αποτελεσματικά νομικά συστήματα κτλ. κτλ. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι λίγο πολύ αυτό είναι ο συμβασμός με τον κύριο Κοφεράτη. Τώρα κατά τα άλλα, τα άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την έκθεση αυτή, μπορούμε να τα συζητήσουμε με τους συναδέρφους και να δούμε αν έχουν κάποια παρατήρηση. Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας και εσάς κύριε Πρόεδρε. Όπως επίσης να συγχαρώ και τον ε, επικεφαλής μας της μονάδας για τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά. Πρόεδρος. Ναι, το είπαμε στην αρχή. Αλλά βέβαια κάποιοι καθυστέρησαν. Όντως έχουμε γενέθλια εδώ και είπαμε τα χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ. Τώρα παρακαλώ κύριε Κοφεράτη. Σκιώδης εισηγητής για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ιδιαίτερε ευχαριστίες οφείλονται στο συνάδελφο Σβάμπ για την διαθεσιμότητά του, για την ετοιμότητά του να μα ακούσει. Ευχαριστίες επίση προς τους άλλου και όδης ε, συζητητέ. Οι συμβιβαστικέ λύσει είναι ικανοποιητικέ. υπήρξαν καρπός ενό κοινού προσανατολισμού. Δυσκολευτήκαμε να βρούμε τι πιο αποτελεσματικέ διατυπώσει για να περάσουμε την ιδέα που όλοι συμμεριζόμασταν και για το λόγο αυτό πιστεύω ότι φτάσαμε σε μια σφαιρική προσέγγιση πολύ θετική και κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη των συναδέλφων μου. Ανοιχτό παραμένει ένα μικρό πρόβλημα. Θα αποφασίσει στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την δική της συλλογική εργασία. Οι συνάδελφοι από το Λαϊκό Κόμμα ομολογώ ότι δεν έχουμε καταλάβει ε, τη στάση της Επιτροπής και ελπίζουμε να μπορέσουμε να την πείσουμε στο μέλλον. Διαφορετικά θα ψηφίσουμε χωριστά. Η... Κατά τα λοιπά, ε, το όργο αυτό έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και εκφράζω την ικανοποίησή μου γι' αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ε, είμαι ευχαριστημένος που υπάρχει υποστήριξη από όλες τις πλευρές. Δεν υπάρχει κανείς από τους κοιόδης εισηγητές ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει το λόγο. Όχι, λοιπόν, ολοκληρώνουμε και αυτό το σημείο. Α, ο κύριος Σβάμπ. Ε, συνεργαστήκαμε πολύ καλά με τον συνάδελφο Κοφεράτη και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και μετά. Τώρα για τις συλλογικές προσφυγές θα ήθελα να προσθέσω το εξής για να το ξεκαθαρίσω. Ε, σε γενικές γραμμές δεν είμαστε κατά στις συλλογικές απαιτήσει αποζημίωσης των καταναλωτών. Ε, ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος είναι αυτό πάνω στο οποίο έχουμε ίσως ξεχωριστή άποψη. Τον Μάρτιο η Επιτροπή θα προτείνει κάποιο σύστημα υλοποίησης και θα δούμε. Θα συνεργαστούμε επικοδομητικά. Να μην δημιουργούμε όμως εσφαλμένες εντυπώσεις, ε, να μην δημιουργούμε εσφαλμένες εντυπώσεις για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Ε, ίσως θα πρέπει να πάμε πέρα από το αμερικανικό σύστημα. Ε, έχουμε κάποιες επιφυλάξεις. Ασφαλώς θα επανέλθουμε στο θέμα των συλλογικών αγωγών. Ευχαριστώ. Μπορώ να προσθέσω κι εγώ ένα σχόλιο. Ο κύριος Χατζημαρκάκης, ο σκιώδης εισηγητής, μόλις μπήκε στην αίθουσα και θα δώσω και σε αυτόν τον λόγο πριν συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή. Χαίρομαι που μπορέσαμε να εργαστούμε από κοινού στην Επιτροπή. Γι' αυτό και υπάρχουν τόσο λίγες τροπολογίες. Τις περισσότερες μπορούμε να τις στηρίξουμε. Ε, μερικές βέβαια παρουσιάζουν κάποιες δυσκολίες, αλλά έχουν ήδη σχολιαστεί. Ο κύριος Βάμπ συγκεκριμένα μας περιέγραψε τις δυσκολίες που υπάρχουν και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Νομίζω όσο αφορά την υλικοτεχνική οργάνωση, η επιτροπολογία 8 νομίζω δεν έχει θέση εκεί. Λίγο έχει παραμεληθεί ε, η έννοια των logistics τα τελευταία χρόνια και οι σχετικές ευρωπαϊκές εταιρείες. Στη συνέχεια για την ε, ενέργεια, η τροπολογία για την ενέργεια, νομίζω διορθώνει τα κακός κείμενα και πρέπει να επιμείνουμε. Καλό θα έχουμε έναν επίτροπο που ανήκει στο ίδιο κόμμα με εσά, που προέρχεται από το ίδιο Μόσπονδο Κρατήδιο της Γερμανίας και που θεωρεί ότι έληξε το θέμα, αλλά δεν ισχύει. Τον είδα στην τηλεόραση δηλαδή και μας είπε ότι το θέμα έκλεισε, έκλεισε, έληξε, πράγμα που δεν ισχύει. Ε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να δημιουργείται περαιτέρω γραφειοκρατία και ότι ε, θα υπερκεράσουμε το στόχο αν ε, προσπαθούμε να είμαστε υπερβολικά προστατευτικοί απέναντι στις εταιρείες. Πάντως θα στηρίξουμε πέραν από την τροπολογία 8 όλες τις άλλες συμβιβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σφάπ, θέλετε να προσθέσετε κάτι, θέλει κάποιος άλλος να λάβει το λόγο πάνω σε αυτό. Όχι. Καλώς λοιπόν. Ε, κλείνουμε τη συζήτηση οριστικά πάνω σε αυτό. Σημείο 16 για αύριο, ε, διαχείριση της εσωτερικής αγοράς. Εισηγητής ο κύριος Σφάμπ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ασφαλώς χαρούμενος που μπορέσαμε να εργαστούμε με τέτοια ταχύτητα. Για άλλη μια φορά, δεν υπάρχει κανείς εκπρόσωπος εδώ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να παρακολουθήσει τη συζήτηση. Ε, α, είσαστε εδώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Α, τέλεια. Εντάξει, τώρα ησύχασα. Γιατί είναι σημαντικό σήμερα να παρευρίσκεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συζήτηση. Γιατί εδώ στην Επιτροπή μας ε, είμαστε ομόφωνοι ως προς τους στόχους που πρέπει να έχει η διαχείριση της ενιαίας αγοράς. Και συμφωνούμε εδώ και με τον κύριο Κοφεράτη. Ε, είδαμε και τις διαδηλώσεις στη Γερμανία. Νομίζω ότι πρέπει να γίνονται σεβαστοί από όλο τον πληθυσμό οι κανόνες που διέπουν την εσωτερική αγορά. Ε, και θα πρέπει όλοι μας να προασπίζουμε τους κανόνες αυτούς. Και δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό παρά μόνο αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, χαρτογραφήσει την κατάσταση που ισχύει ε, στις ευρωπαϊκές χώρες, στα κράτη-μέλη και προτείνει διορθωτικά μέτρα. Ε, στο Στρασβούργο καταλήξαμε σε κάποιες συμβιβαστικές λύσεις, δεν θα τις αναπτύξω όλες, αλλά θα αναφέρω κάποια στοιχεία τα οποία απαιτούν περαιτέρω εμβάθυνση κατά τη γνώμη μου. Καταρχήν, οι συνάδελφοι από την Γκουε και τους σοσιαλιστές θέλουν μια σαφή παραπομπή στο δίκαιο των εργαζομένων. Θέλουν περισσότερο κοινωνικό μέσα σε αυτή την έκθεση. Θέλουν να τονιστεί η κοινωνική πτυχή σε αυτή την έκθεση. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπως ξέρετε, είναι υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων, γιατί αποτελεί το δίκαιο των εργαζομένων αναπόσπαστο κομμάτι μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Και για το λόγο αυτό ευχαριστώ τον κύριο Κοφεράτη γιατί δεν επιθυμεί να τροποποιήσει την νομοθεσία. Αυτά τα δύο στοιχεία για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι πάρα πολύ σημαντικά στο πλαίσιο του ισχύοντος νομικού για το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η ομοιόμορφη υλοποίηση του δικαίου από όλους. Ε, έχουμε τις θεσμικές μας διαδικασίες εδώ, μια διαδικασία συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Έγιναν όλα αυτά και πρέπει τώρα να τηρηθούν και φυσικά πρέπει να σεβαστούμε την περιβαλλοντική και εργασιακή πτυχή του θέματος, αλλά αυτή, αυτός ο σεβασμός δεν θα πρέπει να αποδυναμώσει το θεσμικό μας πλαίσιο. Ε, σεβαστό το, σεβαστά τα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά και το ευρωπαϊκό δίκαιο πρέπει να εφαρμόζεται παντού και τα δικαιώματα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται ομοιόμορφα παντού. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων. Δεν πρέπει να υπάρχουν παρεμβάσεις άλλων τομέων. Εδώ μιλούμε για μια στρατηγική εφαρμογή των κανόνων που υιοθέτησε η επιτροπή μας. Επιτροπή για την εσωτερική αγορά. Τέλος, η Γκουε έχει κάποιο πρόβλημα με τις αιτιολογικές σκέψεις F και V. Ε, ε, συζήτησα με τον κύριο Ντεγιούγκ και κατανοώ ότι η ομάδα του αντιμετωπίζει δυσκολίες ως προς αυτό. Ε, συνάδελφος Μάντερς και ο συνάδελφος Ντεγιούγκ θα ήθελαν να υπάρξει μια προκαταρκτική διεργασία. Κατά τα λοιπά, το παράρτημα παραμένει αμετάβλητο. Είχαμε μια... Και είχαμε και μια συζήτηση με τον Επίτροπο Μπαγνιά για να δούμε αν θα τροποποιήσουμε αυτό το παράρτημα. Φαντάζομαι ότι θα λάβετε κι εσείς θέση πάνω στα διάφορα σημεία. Θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της πρότασης. Η πρόταση αυτή δεν αφορά πολύ συγκεκριμένα θέματα, αφορά περισσότερο στρατηγικά θέματα και την καλή εφαρμογή των νομοθετικών κανόνων. Υπάρχει μια σειρά νομοθετικών βάσεων, νομικών βάσεων, με συγχωρείτε, που απορρέουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Στο σχέδιο έκθεσης εγώ προτείνω για το άρθρο 26 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά αυτό αφορά μόνο το Συμβούλιο. Ε, γιατί εδώ λέει ότι το Συμβούλιο προσδιορίζει τις προϋποθέσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές των σχετικών τομέων. και ιδίως όσο αφορά την κοινωνική πρόοδο. Υπάρχουν εμείς ως βουλευτές και ως νομοθέτες θέλουμε να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Θέλουμε να προσθέσουμε λοιπόν μια νομική βάση Νομίζω ότι πρέπει να επιλέξουμε μάλλον τη νομική βάση του six-pack, παράγραφος 6. Ε, και νομίζω ότι πρέπει να υιοθετήσουμε ένα ψήφισμα στο άρθρο 121 παράγραφος 1 όταν ε, χρειαζόμαστε μια, έναν καλύτερο συντονισμό των ευρωπαϊκών πολιτικών και θα μπορέσουμε να βασίσουμε την απόφασή μας στην παράγραφο 6. Δεν ξέρω αν υπάρχει συμφωνία από την πλευρά της Κομισιόν για αυτή τη νομική βάση. Ίσως να υπάρξει σύγκρουση με το six-pack. Δεν ξέρω εάν ε, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να δώσουμε τη σημασία που θα θέλαμε στην εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τις ε, συνεισφορές τους και τις συμβολές τους. Περαμένω πολλά από την ψηφοφορία. Πιστεύω ότι είχαμε μια καλή συνεργασία και νομίζω ότι στην με την συζήτηση στην Ολομέλεια θα πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό σήμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ για τις εξηγήσεις αυτές. Από ό,τι κατάλαβα, ο συνάδελφος ε, προτείνει για τα κράτη-μέλη κάποιο είδους ε, εξοδικαστική επίλυση. Ο κ. Σκοφεράτη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο, συνάδελφο ο συνάδελφος ε, έκανε μια πολύ σημαντική εργασία και με πολύ ωραίο τρόπο. Συμφωνώ με απο... συμφωνώ με την αφετηρία του. Πρέπει να προσπαθήσουμε ε, να δώσουμε στις ευρωπαϊκές πολιτικές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη σωστή διάσταση της εσωτερικής αγοράς. Γιατί τα θέματα της εσωτερικής αγοράς ε, διαπλέκονται με όλα τα άλλα. Δεν θα πρέπει να περιέλθει το θέμα αυτό στο περιθώριο. Λόγω δομικών περιορισμών. Έχουμε, Έχουμε συζητήσει πάρα πολύ, προσπαθήσαμε να βρούμε κοινέ συμβιβιστικές προτάσεις με πολύ δυσκολία, με πολύ δουλειά, αλλά και με ανοιχτό πνεύμα, με, με μεγάλη διάθεση και το αναγνωρίζω αυτό και στον εισηγητή. Θεωρώ ότι αναφύονται κάποια προβλήματα. Ήθελα να ανταποκριθώ, να απαντήσω μάλλον σε μια παρατήρηση του εισηγητή σε σχέση με τα κοινωνικά δικαιώματα και τα προβλήματα των εργαζομένων. Ιδίω ε, στα προβλήματα που, έχουν τονίσει, που έχει τονίσει με τις τροπολογίες της ΙΓΚΟΕ. Εγώ θεωρώ ότι στο στο θέμα που συζητούμε πρέπει να γίνει παραπομπή σε μία μόνο πλευρά. Η φυσική αναφορά αυτής της Επιτροπής είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες υπό την ιδιότητά τους ως καταναλωτές. Πιστεύω ότι η λύση που επιλέξαμε μπορεί να κάνει αναφορά στα δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, επομένως των πολιτών και υπό την ιδιότητά τους ως εργαζομένων. Ο πολίτης θα πρέπει να είναι το κυρίαρχο υποκείμενο υπό οποιαδήποτε ιδιότητά του. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια αναφορά, μια παραπομπή, αδιακρίτως αν επιτραπεί η χρήση αυτού του όρου, αδιακρίτως στα δικαιώματα όλων. Ε, αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική πτυχή όσο αφορά τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση της εσωτερικής αγοράς. Για το λόγο αυτό, ίσως θα ε, μπορεί να γίνει λίγο κάποια συμπληρωματική εργασία, έτσι με θετικό πρόσημο. Θα ήθελα να, ζητή, να ρωτήσω τον εισηγητή πώς, βλέ... πώς, θα έβλεπε κάποιες τροπολο... πώς θα έβλεπε τις τροπολογίες που υπέβαλα εγώ για το ευρωπαϊκό εξάμεινο. La proposta che lui fatto. No. Ε, ίσως θα μπορούσε να εξετάσει έτσι ξεχωριστά ο εισηγητής αυτές τις τροπολογίες. Ε, Ευχαριστώ για την Άλντε, τους φιλελεύθερους, δεν υπάρχει κανείς. Άντερ ε, για τους πράσινους. Ναι, θα είμαι αρκετά σύντομη. Συμφωνώ αρκετά με τον κύριο Κομφεράτη και πιστεύω ο, η οριοθέτηση που διάλεξε ο εισηγητής είναι αρκετά ικανοποιητική και εμείς σκεφτήκαμε αρκετά γιατί δεν λαμβάνουμε υπόψη το περιβάλλον, την αηφορία, αλλά εδώ πρόκειται για εφαρμογή. Δεν πρόκειται για την σύνταξη της νομοθεσίας, αλλά για την υλοποίηση, την εφαρμογή, την επιβολή της νομοθεσίας. Και είναι αλήθεια ότι αυτές οι παρατηρήσεις μπορούν να παίξουν ένα ρόλο ε, για να δούμε τι γίνεται με την ε, βιωσιμότητα, τη διατηρησιμότητα. Αυτό θα πρέπει να εμφανίζεται στα διάφορα κριτήρια. Αλλά όταν έχουμε την νομοθεσία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη και σε αυτό το επίπεδο έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Δεν θα πρέπει να ανοίγουμε νέες και για τον λόγο αυτό. Πιστεύω ότι το αίτημα της Γκουε δεν είναι βάσιμο, δεν είναι αιτιολογημένο. Νομίζω στο σημείο Β γίνεται λόγος για συστήματα προειδοποίησης αποτελεσματικά. Θα μπορούσαμε να εργαστούμε με τον τρόπο αυτό νωρίτερο, αλλά θα πρέπει η Επιτροπή να μπορεί να υιοθετήσει ορισμένα μέτρα ή αλλιώ δεν θα υπάρχει συνεκτικότητα. Ο κύριος Ντεγιόγκ δυστυχώς δεν είναι εδώ παρόν, ούτως ή άλλως θα μιλήσω ακόμη μαζί του και στο επίπεδο αυτό νομίζω ότι η λύση αυτή δεν είναι ορθή και για τα υπόλοιπα υποστηρίζω τον εισηγητή και ελπίζω ότι η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις προτάσεις του και περιμένω με ενδιαφέρον τη συζήτηση με τον κύριο Μπαρνιέ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Μακλάρκιν για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ε, ε, έχουμε τους συμβιβασμούς για την σημαντική εισήγηση και το γενικό πνεύμα καλύπτει και τις δικές μου τροπολογίες. Δεν θα ήθελα να ξοδέψω ε, πολύ χρόνο και είχαμε την περασμένη εβδομάδα μια συνεδρίαση για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου για τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Η μόνη ερώτηση που έχω είναι σε σχέση με την συμβιβαστική λύση 5 και ο εισηγητής ζητάει την εισαγωγή της ενιαίας αγοράς στο πρώτο ήμιση το, της συμβιβασμού δεν, δεν ξέρω πολύ καλά τι είναι αυτό το οριζόντιο μέτρο που προτείνει στο δεύτερο μέρος και ποιος, ποια, ποιος είναι ο συλλογισμός ο υποκείμενος αν πρέπει να μην ενώ η αναθεώρηση της ε, οδηγίας πρέπει να θεωρηθεί για να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής, να περιλαφθούν άλλοι τομείς. Ένα οριζόντιο ε, μέσο θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό όταν θα έχουμε ε, το σχέδιο νόμου κλπ και για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε τοπικό επίπεδο. Στην, δεν ήμουνα στην προηγούμενη συνεδρία, ήταν ο εισηγητής αναφέρθηκαν ορισμένα θέματα σε σχέση με ορισμένε τροπολογίε, και θα ήθελα να διευκρινίσουμε ορισμένε αιτιολογήσει για την τροπολογία 14 για την σύσταση 5. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την πρόοδο ε, στην εφαρμογή των εθνικών σχεδίων δράση. και θα πρέπει η Κομισιόν να λάβει όλες τι απαιτούμενε αναγκαίε πληροφορίε για να αξιολογήσει την πρόοδο και εδώ διέγραψα κάτι, διότι θα πρέπει νομίζω τα κράτη-μέλη να παρακολουθούν, να επιτηρούν τα δικά τους σχέδια δράσης σε συνεργασία με την Επιτροπή. Νομίζω ότι η διατύπωση αυτή, η σύσταση από τον εισηγητή είναι κάπως δυνατή η διατύπωση, αν θα μπορούσαμε να δούμε αυτή τη διατύπωση για την τροπολογία 119 για την διαγραφή της σύστασης 6 σύσταση στα κράτη-μέλη και θα πρέπει η Επιτροπή να έχει τα μέσα για, που προβλέπονται από την συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε σε μια σύσταση άρθρα από τη συνθήκη. Ε, εδώ θα πρέπει ο εισηγητής να μου δώσει την άποψή του για το θέμα αυτό και για, το 100, για την 125 και πάλι διέγραψα ε, ένα, κάτι από την σύσταση 7F σχετικά με τη σύσταση στα κράτη-μέλη βάσει πρότασης από την Κομισιό. Νομίζω ότι νομίζω πρέπει να βάλουμε το βάρος, να ρίξουμε το βάρος στο Συμβούλιο που κάνει συστάσεις στα κράτη-μέλη σχετικά με τις προτεραιότητες και αυτά έχουν γίνει. Θα ήταν καλό να ίσως να προσθέσουμε κάτι άλλο, αλλά και πάλι εκτιμώ τις απόψεις του εισηγητή. Έχουμε όλοι τις ίδιες προτεραιότητες Ίσως ο τρόπος που τις εκφράζουμε είναι διαφορετικός, γι' αυτό θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι εστιάζονται σε αυτό που θέλουμε και ότι δεν δημιουργούν ε, περισσότερο φόρτο. Θα, ε, ε συμφωνώ με τον εισηγητή για την ανάγκη να αποφύγουμε να εστιαζόμαστε στα κοινωνικά δικαιώματα και να εστιαστούμε πολύ περισσότερο στην εφαρμογή όσον αφορά στο φάκελο αυτό. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω άλλο σκιώδη συγητή. Δεν ξέρω αν υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν να λάβουν το λόγο. Δεν νομίζω. Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία την παρέμβαση της Επιτροπής. Δεν ξέρω ποιος θα λάβει το λόγο στο όνομα της Επιτροπής. Πολύ καλά. Ο κύριος Βάμπ θα απαντήσει μόνος του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για τις συνεισφορές τους, οι, οποίοι, οι οποίες συνέβαλαν όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Θα ήθελα να αρχίσοντας να σας πω ότι ότι μπορεί αυτό να είναι ε, χρήσιμο για να διευκρινίσουμε τα πράγματα ως προς το στόχο του κειμένου, όπως ο κύριος Κομφεράτη το είπε, θα μπορούσαμε ίσως εδώ να επιμείνουμε πάνω στο γεγονός ότι δεν ε, υπάρχουν ε, μόνο οι προσδοκίες ε, οι κρατικές, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα να έχουμε ενιαία εφαρμογή, αλλά όλοι θα πρέπει να αισθανθούν ότι είναι ενδιαφερόμενοι. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κάτι να έχει υπάρχει μια καλύτερη διακυβέρνηση στο επίπεδο της εσωτερικής αγοράς, διότι σκεφτόμαστε τους εργαζόμενους, άνδρες και γυναίκες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι αυτό το οποίο επιθυμούμε είναι να λάβουμε υπόψη ε, τους εργαζόμενους, ε, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι είναι και καταναλωτές και καταναλώτριες. Θα πρέπει να τονίσουμε κυρίως και να δώσουμε έμφαση στην εφαρμογή, στην επιβολή και αυτό είναι κάτι σημαντικό για τις διάφορες πολιτικές ομάδες όπως και για τη δική μου την πολιτική ομάδα το έχουμε ήδη πει αυτό και καμιά φορά είναι πλεονασμός να επιμένουμε πάνω σε τέτοια σημεία το ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε μια προφορική τροπολογία για το θέμα αυτό. για τις άλλες τροπολογίες οι οποίες αναφέρθηκαν από τον συνάδελφο Κομφεράτη για το Six Pack. Συμφωνώ πλήρως μαζί σας και ακόμη και αν πρόκειται για στοιχεία τα οποία δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα, πρόκειται εδώ μάλλον για ένα θέμα πολύ περισσότερο λογοτεχνικό παρά πολιτικό. Η κυρία Ρόλ, βεβαίως θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας και θα ήταν καλό αν μπορούσαμε να πείσουμε τον συνάδελφο De Jong της Γκουε να υιοθετήσει την άποψή μας, διότι υπάρχει μια διχογνωμία στο επίπεδο αυτό. Κυρία Μακλάρκινγκ, αναφερθήκατε σε μια τροπολογία, κυρίως την τροπολογία 114, στο επίπεδο αυτό. Θα ήθελα βέβαια πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την ομάδα σας για την υποστήριξή της, αλλά έχετε δίκιο από την άποψη αυτή το κείμενο δεν είναι αρκετά κρυβές. Δεν είναι για έλλειψη διπλωματίας, είναι... αλλά θέλουμε να έχουμε σαφέστερο κείμενο. Όπως κατέδειξε η συζήτηση, δεν είναι πάντοτε εύκολο να είμαστε αρκετά κρυβείς αν θέλουμε τα όσα υιοθετούνται, υιοθετηθούν, να εφαρμοστούν δεόντως και να αποφύγουμε κάθε παρεξήγηση. Είναι σημαντικό να νομοθετούμε ορθώς, καλά και θα πρέπει να καλύψουμε ορισμένες ελλείψεις σε αυτό το επίπεδο. Αν θέλουμε όλα να τελεσφορήσουν καλά, θα πρέπει να δούμε πώς με τα κράτη-μέλη θα υλοποιήσουμε τα πράγματα με τον καταλληλότερο τρόπο. Κρίμα που δεν υπάρχει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λαμβάνει τον λόγο. Δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο να αναφέρω τις άλλες τροπολογίες τη μία μετά την άλλη. Νομίζω ότι συμφωνούμε ως προς την ουσία το περιεχόμενο. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι τροπολογίες που θα προταθούν από τις άλλες ομάδες και του χρόνου. Βάσει όλων αυτών των τροπολογιών θα δούμε τι μπορεί να γίνει για να παραμείνει λογική εισήγησή μας και μετά, η συζητή, με, μετά τις συζητήσεις με τον Επίτροπο Μπαχνιέ θα δούμε ποια είναι σαφώς η θέση της Επιτροπής και αυτό που είναι σημαντικό για όλους και για την Κομισιό και για μας είναι για την ώρα η Κομισιό δεν έχει τα κατάλληλα μέσα και εργαλεία ούτω, ώστε οι προσαναταλισμοί αυτοί να ληφθούν καλά υπόψη. Η κυρία Γκέπχαρτ το είπε καλά για μια ολόκληρη σειρά εισηγήσεων υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία εμείς αγνοούμε και είναι δύσκολο να δούμε σαφώς τα πράγματα και το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να εξακολουθήσουμε να ασκούμε πίεση πάνω στην Κομισιό για να συνεχιστούν τα πράγματα και για να μπορέσουμε να προδώσουμε ακόμα περισσότερο, να αναλάβουμε περισσότερη ευθύνη και έχουμε την εντύπωση ότι τα πράγματα, τα θέματα που εκκρεμούν θα μπορέσουν να αποτελέσουν αντικείμενο συμβιβασμού του χρόνου. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ που αναφερθήκατε σε αυτό το σημαντικό θέμα. Η Κομισιό είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και για τον έλεγχο, αλλά να στα κράτη-μέλη να δουν πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά. Είναι αρμόδια τα κράτη-μέλη και υπεύθυνα στη συνθήκη της Λισαβόνας το βλέπουμε είναι καλή εμπιστοσύνη αλλά και ο έλεγχος είναι ακόμη καλύτερος και η Κομισιόν βεβαίως είναι για μας σημαντικός προσκεκλημένος βεβαίως ε, τροποποιήθηκε σημαντικά η μερίσια διάταξη ίσως γι' αυτό δεν υπάρχει κανείς από πλευρά της Κομισιόν διότι αυτή η ανακοίνωση κοινοποιήθηκε αρκετά αργά. Ε, περνάμε τώρα στο σημείο 7 ε, μια νέα ατζέντα για την ευρωπαϊκή πολιτική ε, καταναλωτών. Δίνω τον λόγο στον Ιζέντε Μικουέλ Γκάρθες Ραμόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να λάβω τον λόγο σε σχέση με το σχέδιο έκθεσης που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή για μια νέα ατζέντα για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σας πω ευθύ εξ αρχής ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που χρήζει εξέτασης περαιτέρω και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας θα πρέπει να συντάξουμε μια έκθεση η οποία θα είναι η καταλληλότερη και η ορθότερη. Θα αρχίσω ευχαριστώντας την Επιτροπή για την πρωτοβουλία της και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Επιτροπή Περιφερειών και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ε, για την αποφασιστικότητα, για το ψήφισμα και την γνωμοδότηση και να ευχαριστήσω ορισμένες οργανώσεις και ενώσεις καταναλωτών που με υποστήριξαν για τη σύνταξη της εισήγησής μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ειδικού επίσης από την Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από την πολιτική ομάδα που με στήριξαν προς αυτή την κατεύθυνση. Το σχέδιο που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει διάφορες πρωτοβουλίες για τους καταναλωτές για την περίοδο 2014 με 2020. Άρα λοιπόν περνάμε από το βραχυπρόθεσμο στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο. Και εδώ βλέπουμε να αναφέρονται διάφοροι στόχοι, διάφορες προκλήσεις πιο σωστά, πολύ σημαντικές. Και θα αρχίσω από την διαδικασία παγκοσμιοποίησης των αγορών. και την ε, δημοσιονομική απορρίθμιση. Και θα αναφερθώ επίσης και στην κύρανση του πληθυσμού. Αυτές είναι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε οπωσδήποτε. Είναι προκλήσεις και για τους καταναλωτές, οι οποίοι διαπιστώνουν το χάσμα ανάμεσα στο ε, εθνικό διαδικτυακό εμπόριο και το διασυνοριακό μεγαλώνει. Βλέπουμε επίσης να αυξάνεται η ανησυχία των καταναλωτών όσον αφορά τα τρόφιμα, την ασφάλεια των τροφίμων. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε 8 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη που δεν μπορούν να επιτρέψουν στους εαυτούς τους να έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά, βασικά για τη ζωή τους. Όλοι αυτοί οι στόχοι και όλες αυτές οι προκλήσεις λοιπόν μας υποχρεώνουν να καταλήξουμε σε κάποιες προτεραιότητες και αυτό ακριβώς είναι και το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους καταναλωτές. Εκεί λοιπόν περιλαμβάνουμε την υγεία, την ενέργεια, τα ασφαλή τρόφιμα, την ψηφιακή τεχνολογία, την μείωση των ανισοτήτων, την πρόθεση μιας οικονομίας με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και επίσης ένα άλλο στοιχείο είναι η προσοχή που πρέπει να δώσουμε στις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας μας, παιδιά κλπ. Υπάρχουν διάφορες ανάγκες στα πλαίσια αυτά. Μέσα από κατάστασης, για παράδειγμα, στήριξη οργανώσεων καταναλωτών που να χρηματοδοτούνται επαρκώς, διάφανες διαδικασίες, την ε, διαπαιδαγώγηση των καταναλωτών και ένα μητρό καταναλωτών ώστε εκεί να συμπεριλαμβάνονται όλες οι ευρωπαϊκές οργανώσεις που ασχολούνται με τους καταναλωτές. Αυτά θα έλεγα σε μια πρώτη μου παρέμβαση είναι τα στοιχεία κλειδί που καταλήγουν σε 18 προτάσεις που περιλαμβάνω στην έκθεσή μου και που δεν θα σας τα επαναλάβω, είναι αυτά που σας είπα λίγο πολύ μέχρι τώρα. Απλώς να σας πω ότι το επίπεδο ε, εφαρμογής πρέπει να είναι το ίδιο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι οι στόχοι και οι προκλήσεις πρέπει να εξετάζονται από πλευράς του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου που θέλουμε να έχουμε. Όπως επίσης και η εποπτεία, ο έλεγχος της αγοράς πρέπει να είναι πράγματα που γίνονται με αποτελεσματικούς μηχανισμούς, όπως και επίλυση διαφορών. Τα συστήματα online διευθέτησης διαφορών να υπάρχουν ή οι συλλογικές προσφυγές να αποτελούν μέρος οπωσδήποτε της ε, πολιτικής μας στρατηγικής υπέρ των καταναλωτών. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ραμόν, ήμουνα με την κυρία Ρέντινγκ, όπως είπα και πριν. Θέλω να ευχαριστήσω και όσους ήρθαν ε, στο μεταξύ κατά την διάρκεια που έλειπα εγώ, την κυρία Κέπαρτ για παράδειγμα και λοιπόν. Λοιπόν, ε, κύριε Σβάμπ, εσείς θα μιλήσετε εκ μέρους του ΕΛΚ. Όχι εκ μέρου τη κυρία Ρέντινγκ πάντως, ε. μην τα μπερδεύετε. Πρώτον, τα σχόλιά μου έχουν να κάνουν πρώτον με τα γενικά σχόλια και τα λέω εκ μέρους του κύριου Κανιέτη, ο οποίος ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Της, κύριε Κανιέτη, η οποία μου είπε πρώτα απ' όλα ότι εκείνη και το ΕΛΚ θεωρούμε ότι είναι θετικά τα όσα αναφέρει ο εισηγητής για την προστασία των καταναλωτών. Οι περισσότερες από τις προτάσεις του μας ε, βρίσκουν σύμφωνους σε εμάς από το ΕΛΚ. Όμως, λέει ότι οι ευκαιρίες για την απασχόληση και οικονομική ανάπτυξη είναι πράγματα που θα πετύχουμε αν φροντίσουμε τις επιχειρήσεις μας. Άρα η έκθεση αυτή δεν πρέπει να είναι κατά των επιχειρήσεων, γιατί τότε θα στείλουμε λάθος μήνυμα στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι κι αλλιώς είχαμε πάει μαζί στις Ηνωμένε Πολιτείες και το ξέρει και ο συγκεκριτής πολύ καλά. Τώρα εξαιτία τη σημερινή κατάσταση τη οικονομία από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε τον ιδιωτικό τομέα με επιπλέον κόστο. Και η κυρία Κανιώτε λέει ότι η τελική εκδοχή της έκθεσης να βοηθήσει με ιδέες υπέρ του διασυνοριακού ε, εμπορίου και να ενισχυθεί η πτυχή B2C. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα σχόλια που έχω να κάνω εγώ από τη δικιά μου την πλευρά προσωπικά. Αλλά προηγουμένως όταν αναφέρθηκα σε αφιβολίες το απίθυνε προς τον κύριο Κοφεράτη για το γιατί το ΕΛΚΑ δεν είναι τόσο θετικό όσον αφορά τις συλλογικές προσφυγές όπως οι άλλες ομάδες, να σας εξηγήσω. Εμείς ξεκινάμε από την αρχή που λέω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας κάνει μια πρόταση, ιδιαίτερα για το private enforcement και τους γενικούς κανόνες. Δεν είμαστε κατά της εφαρμογής αυτής για τις συλλογικέ προσφυγές. Απλώς η νομική κωδικοποίηση φαίνεται να είναι πιο δύσκολη Γι' αυτό και είμαστε κάπως επιφυλακτικοί. Όσον αφορά τώρα το σημείο σιγματάφ, το F, σας παρακαλώ να δείξετε κάποια επίκαια. Έρχομαι τώρα στο H, ήτα. Εδώ, όντως η ελευθέρωση αυτή καθεαυτή δεν βοήθησε ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους πολίτες. Αλλά η ελευθέρωση, αν μη τι άλλο, οδήγησε σε κάποιες επιμέρους βελτιώσεις, όπως στην διασφάλιση κάποιων θέσεων απασχόλησης. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε ότι το ΙΤΑ είναι κάπως ε, μονομερές. Έπειτα εκεί που αναφέρεται Ε, το γεγονός ότι στην Ισπανία, για παράδειγμα, διώχνουν από τα σπίτια τους τους ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν, όντως είναι κάτι τραγικό για τους καταναλωτές. Από την άλλη, δεν μπορούμε εμείς εδώ να δώσουμε την εντύπωση ότι αυτό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Όχι, γιατί έχει να κάνει με την κατάσταση στην Ισπανία. Πάντως το καταλαβαίνω ότι για τους ανθρώπους εκεί είναι τραγικό. Συμφωνούμε επίσης για το ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει πολύ μεγάλη σημασία και συμφωνούμε και πολλές άλλες προτάσεις του εισηγητή. Σας ευχαριστούμε για την έκθεσή σας και περιμένουμε τη συνέχεια της συζήτησης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ροσφόρ. Πρόεδρε, κύριε εισηγητά, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα συγγνώμη που καθυστέρησα, ήμουν στο γραφείο μου και δούλευα και ε, δεν είχα καταλάβει ότι είχε προχωρήσει τόσο πολύ η ημερήσια διάταξη. Συγγνώμη που ήρθα τόσο αργά. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γαρσές Ραμόν για την ε, έκθεσή του αυτή που είναι τόσο ενδιαφέρουσα και ευχαριστώ πολύ επί τη ευκαιρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υπέβαλε το θεματολόγιο αυτό, ένα ευρωπαϊκό θεματολόγιο, μέσα στο οποίο βλέπω να συμπεριλαμβάνονται πολλές από τις ανησυχίες μου. Σήμερα ε, μιλούσαμε για... Ε, μιλάμε μάλλον για το θεματολόγιο για τους καταναλωτές. Πριν από λίγο καιρό μιλούσαμε για την ατζέντα για τους καταναλωτές. Ε, η ορολογία αλλάζει. Πάντως πολλά σημεία στην έκθεση Γκαρσία Ραμών με βρίσκουν σύμφωνο. Ίσως δεν είναι αναγκαίο εδώ να τα απαριθμίσω, μια που συμφωνώ, όμως υπάρχουν κάποια στοιχεία για τα οποία θέλω να πω ήδη από σήμερα το βράδυ ότι η ομάδα μου έχει κάποιες επιφυλάξεις. Κάποια εξάλλου από τα σημεία αυτά τα ανέφερε και ο συνάδελφος Ανδρέας Σφάπ. Κάποια από αυτά έχουν επιστήσει την προσοχή μας, το ίδιο δηλαδή όπως συνέβη και με τον Ανδρέα. Αυτό όμως που εγώ θέλω να πω εδώ για το στυλ της έκθεσης είναι ότι σε κάποιες στιγμές δημιουργείται μια πολεμική που δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητη για ένα τέτοιο θέμα. Στην Επιτροπή μας και τα προηγούμενα χρόνια προσπαθούσαμε πάντα να καταλήξουμε σε συνενέσεις, σε συνενετική δουλειά βελτιώνοντας, ε, καταλήγοντας σε συμβιβασμούς. Πάντα καταφέρναμε ένα καλό αποτέλεσμα. Θα μιλήσω κι εγώ, όπως και ο Ανδρέας Σφαμπ, για τις διάφορες παραγράφους εδώ, με τη σειρά λίγο πολύ. Πρώτα απ' όλα, η πρόταση που γίνεται στην παράγραφο 3 για να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό μητρό ενώσεων το οποίο θα διευκολύνει το σχηματισμό ευρωπαϊκών ενώσεων. Εγώ δεν είμαι πεπισμένο ότι έτσι πρέπει να γίνει. Και ρωτάω τον εισηγητή, η διατύπωση ως έχει στην παράγραφο 3 για μένα είναι ασαφή. γενική, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. Φυσικά και θέλουμε να στηρίξουμε και εμείς τις ενώσεις υπέρ των καταναλωτών. Φυσικά και συμφωνούμε να υπάρξει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να δημιουργηθούν δίκτυα τέτοιων ενώσεων, αλλά το μητρό στο οποίο αναφέρεστε δεν μου αρέσει τόσο πολύ και δεν ξέρω και τι ακριβώς εννοείται με αυτό. Παράγραφος 4. Συμφωνώ με τον εισηγητή και του το λέω. Αυτή η διαβίου κατάρτιση με βρίσκει σύμφωνο. Συμφωνώ ότι αρχίζει από το σχολείο, είναι κάτι μόνιμο και ακριβώς γι' αυτό δεν πρέπει να σταματάει στο σχολείο. Εδώ λέτε ότι ξεκινάει από το σχολείο. Ζητάμε από το σχολείο πάρα πολλά πράγματα. Το σχολείο όμω δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Παράγραφος 6 ενιαίοι κανόνες για την ε, εξασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων. Συμφωνώ. Αλλά θέλω να επιμείνω στο θέμα της ε, της, ε, του να βρούμε από πού προέρχεται το προϊόν, η χνηλασιμότητα του προϊόντος. Αυτό είναι πολύ βασικό. Έπειτα και το ηλεκτρονικό εμπόριο, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε για το ότι πρέπει να είναι ηθικό το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σίγουρα πολλά έχουν να γίνουν ακόμα για να το πετύχουμε αυτό. Έχουν γίνει και κάποια πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει καταδείξει τις ελλείψεις Δύο λόγια τώρα και στις παραγράφους 8 και 10. Κατάλαβα ότι ο Καντρέα Σιβάπ λίγο πολύ το ίδιο λέει, με αυτό θέλω να πω και εγώ για την παράγραφο 8. Πρέπει να δίνουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Εδώ. Ακόμα και εγώ εννοείται ότι είμαι υπέρ των καταναλωτών και νιώθω απόλυτα αλληλέγγυος απέναντί τους για τις υποθήκες τους και τα λοιπά. Οι υποθήκες όμως δεν είναι απαραίτητα ένα ξεκάθαρο προϊόν καταναλωτικό. Είναι μια χρηματοπιστωτική υπηρεσία για τους καταναλωτές. Καταναλωτές οι οποίοι μάλιστα είναι οικονομικοί φορείς στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι οποίοι αποκτούν το σπίτι τους εφόσον όλα πάνε καλά. Οπότε να μην βάζουμε ονόματα. Έπειτα για τους ευάλωτους ε, καταναλωτές. Γιατί ο εισηγητή μα προτείνει εδώ να αναφέρουμε συγκεκριμένα τις μεταφορές σε σχέση με τους ευάλωτους καταναλωτές. Αφού θέλετε να είμαστε συγκεκριμένοι, εγώ συμφωνώ να συγκρίνουμε τις τιμές. Γι' αυτό και στο θεματολόγιο για τους καταναλωτές συμφωνώ ότι αναφέρεται πολύ γενικά. Να διευκρινιστεί περισσότερο παρακαλώ. Τελειώνω. Παράγραφος 15 για την πρόταση της ε, νομικής αρρωγής και δικαστικής αρρωγής για, δωρεάν για τους άνεργους. Εδώ προτείνεται ένας μηχανισμός, ο οποίος δεν ξέρω κατά πόσο συντονίζεται καλά και διατυπώνεται καλά σε σχέση με το τι λέμε σε άλλα κείμενα που έχουμε μελετήσει εδώ στην Επιτροπή μας, κυρίως για τις εναλλακτικέ μορφές ε, διακανονισμών, επίλυσης διαφορών. Εδώ νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ, δεν συντονίζεται καλά με ό,τι άλλο κάνουμε εδώ στην Επιτροπή μας για το ίδιο θέμα. Τέλος να σας πω και κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ ε, και που είπε ο Αντρέας Σβάμπ, δεν συμφωνώ με τον Αντρέα Σβάμπ δηλαδή. Το έχω πει ξανά και ξανά εδώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό βέβαια να υπάρχουν συλλογικέ προσφυγέ. Πάντως για άλλη μια φορά εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα μιλά για αυτό το θέμα πολύ γενικά, για την ευρωπαϊκή προσέγγιση, τι εναλλακτικέ κτλ. Καλό θα ήταν να είναι πιο συγκεκριμένη. Στο πρόγραμμα εργασίας για το 2013 φοβάμαι ότι για αυτές τις λογικές προσφυγές δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Αλλά εμείς αυτή την εποχή θέλουμε να εγκρίνουμε ε, αυτά τα θέματα που έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία ε, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης ενιαίας πράξης. Οπότε, αν θέλουμε να συμπληρωθεί αυτή η εσωτερική αγορά, πρέπει να έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Άρα, κάποιες, ε, έτσι, κάποια χτενίσματα πρέπει να γίνουν για να είναι καλύτερα ισορροπημένο το κείμενο. Ε, πρώτον και δεύτερον να ληφθούν υπόψη παρατηρήσεις μου για το ευρωπαϊκό θεματολόγιο και να προσθεθεί το θέμα της σύγκρισης των τιμών. Εκεί να πάμε πιο μακριά από ό,τι αναφέρει το κείμενο του εισηγητή. Αυτά, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν όλοι τόσο πιο σύντομη πριν έρθετε, γι' αυτό προχώρησε τόσο ημερήσια διάταξη όπως λέτε. Λυπάμαι γι' αυτό. Η κυρία Ρούλε είναι η επόμενη από τους σκιώδες εισηγητές και μετά κι εγώ είμαι σκιώδης, οπότε μετά θα πάρω εγώ τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να σας μεταφέρω κάποιες παρατηρήσεις μου. Πρώτα απ' όλα, στο σημείο G, θέλω να διευκρινίσουμε κάποια σημεία. Λέει ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τις χρηματοπιστωτικές αγορές και υπηρεσίες ή καταναλωτές. Πολύ ωραία. Και το δεύτερο όμω κομμάτι, εκεί που μιλάτε για την κεντρική τράπεζα και για τον ρόλο του επιδιαιτητή, εδώ δεν νομίζω ότι είναι καθήκον τη δικιά μα επιτροπή να αναφερθεί σε αυτά. Εμεί πρέπει να επιμένουμε περισσότερο στην ενημέρωση των καταναλωτών. Εκεί είναι που υπάρχουν ελλείψει. πώ δηλαδή να ενημερώνεται καλύτερο ο καταναλωτή για τι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίε, πώ θα υπάρχει διαφάνεια και όσον αφορά και το κόστο των συμβουλών αυτών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Σημείο 8. Για μένα υπάρχει κάτι που δεν είναι αρκετά σαφές εδώ. Δεν βλέπω τελικά τι ακριβώς θέλει ο εισηγητής. Σημείο 6 επίσης. Η ασφάλεια τροφίμων. Η ασφάλεια προϊόντων. Πρέπει να μιλήσουμε εδώ για την εποπτεία της αγοράς. Η κυρία Σάλντε Μόζε εδώ και χρόνια το ζητάει αυτό. Κάποια στιγμή ανακοινώθηκε, αλλά εδώ νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε και να μπει. Η εποπτεία των αγορών δηλαδή. Καλό θα κάνει, κακό δεν θα κάνει να το έχουμε στο σημείο 6. Σημείο 13 τώρα. Από ό,τι καταλαβαίνω εδώ τίθεται θέμα ε, λιανικών ε, πωλήσεων. Έτσι δεν είναι εμπορία λιανική προϊόντων. Η κυρία Κορέτσα Βίλτ έχει κάνει αρκετά πράγματα εδώ. Έχουμε ένα καλό σημείο εκκίνησης. Δεν πάμε αρκετά μακριά, αλλά τουλάχιστον α λάβουμε υπόψη μα αυτά που λέει εκείνη. Δεν χρειάζεται να υπάρχει επικάλυψη στη δουλειά μα. Ευχαριστώ. σε ευχαριστούμε πολύ. Να κάνω κι εγώ κάποια σχόλια τώρα, μια που είμαι κι εγώ σκιώδη. Συμφωνώ με τους συναδέρφους που είπαν αυτό που θα σας πω κι εγώ. Μην ξεχνάμε ποιο είναι το θέμα μας. Έτσι, σχολιάζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τους καταναλωτές. Όταν διάβασα λοιπόν αυτή την έκθεση για πρώτη φορά, τι μου έκανε εντύπωση. Η δουλειά που κάνουμε, δεν βλέπω γιατί δεν χρειάζονται πέντε σελίδες. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν δύο σελίδες ε, συστάσεων. Και θέλω, επιτρέψτε μου να το πω στον εισηγητή, γιατί εκείνος θα μας κάνει προτάσεις τελικά. Στην αιτιολογική του έκθεση υπάρχουν διάφορα σημεία τα οποία δεν έχω στι προτάσει. Στην πρώτη παράγραφο, για παράδειγμα, λέει ότι πρόκειται για μια φιλόδοξη προσέγγιση και ζητάει από την Επιτροπή να συντάξει επίση πράσινη βίβλο για του Ευρωπαίου καταναλωτέ, που θα είναι προ όφελο των οργανώσεων προστασία των δικαιωμάτων καταναλωτών, των πολιτών και των εθνικών κοινοβουλίων και κυβερνήσεων. Αυτό θα ήθελα να το δω στι συστάσει του εισηγητή και δεν το βλέπω εκεί. Η αποτελεσματικότητα της έκθεσης θα ενισχυθεί εφόσον εμείς τονίσουμε πράγματα για τα οποία είμαστε εμείς αρμόδιοι. Υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία εδώ. Πάντως, υπενθυμίζω στον εισηγητή ότι εμεί δεν είμαστε υπεύθυνοι ούτε για του κινδύνου από τις νέες τεχνολογίες ούτε για την ασφάλεια τροφίμων. Αυτά δεν είναι δικά μας θέματα. Εντάξει, μπορούμε να τα σχολιάσουμε, αλλά μέσα σε κάποιο πλαίσιο, έτσι. Ούτε είμαστε υπεύθυνοι για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ούτε είμαστε υπεύθυνη για τη συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια, την φορολογία κτλ. Στην πράξη, λοιπόν, δεν ξέρω αν τελικά για μας ή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι για να περιληφθεί στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο του καταναλωτέ Ίσως ο θα πρέπει να συναντηθεί με τους ε, σκιώδεις εισηγητές και να εξετάσει καλύτερα το προφίλ. Τελικά τι θα έπρεπε να μπει στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο από εμά. έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις μελλοντικέ επίσης ανάγκες των καταναλωτών. Αυτά που λέτε για το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι πολύ σημαντικό. Η εφαρμογή όμως των κεκτημένων, των ήδη κεκτημένων για τον καταναλωτή είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα Υπάρχουν δικαιώματα των καταναλωτών που υπάρχουν μέσα στα όσα έχουμε αποφασίσει μέχρι τώρα, που όμως δεν εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες μέλη και δεν υπάρχουν και μηχανισμοί επιβολής. Τα περί κατάρτισης είναι επίσης πολύ σημαντικά που λέτε. Και επίσης νομίζω ότι έχετε δίκιο στην αιτιολική σας έκθεση που επικεντρώνεστε στο βαθμολόγιο των καταναλωτών όσον αφορά τις επιδόσεις. Πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία όντως να τα δούμε αυτά, γιατί έχουμε κάνει χωριστή έκθεση, αλλά το γεγονός ότι οι καταναλωτές πολλές φορές δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και ότι πρέπει να υπάρξει διαπαιδαγώγηση των καταναλωτών, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό ίσως να το δούμε περισσότερο σε βάθος, να δούμε δηλαδή τι θα μπορούσε σχετικά με αυτό να συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο. Βρίσκω λοιπόν ότι είναι πολύ χρήσιμο το πλαίσιο που θέτεται, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μπείτε πιο πολύ στις λεπτομέρειες. Λοιπόν, ε, χαίρομαι που βλέπω εδώ την κυρία Μάντων, αλλά πρέπει να πω ότι προχωρήσαμε πολύ γρήγορα. Τι να κάνουμε, συγγνώμη γι' αυτό. Η κυρία Κέπαρτ όμως θέλει επίσης το λόγο, έτσι δεν είναι. Παρακαλώ, κυρία Γέπαρτ. Ή όχι. Ή κυρία Γέπαρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτό το πολύ καλό σχέδιο έκθεσης. Άκουσα με προσοχή αυτά που είπατε, κύριε Πρόεδρε. Είστε μάλλον πιο ενημέρος από εμένα έχουμε πολύ περιορισμένο χώρο. Ε, η αιτιολογική έκθεση δεν μπορεί να τροποποιηθεί πλέον. Μπορούν όμως να υπάρξουν ε, τροπολογίες εκ μέρους του εισηγητή. Δεν θα ήθελα να ξαναρχίσω τις επικρίσεις, αλλά κάποια στοιχεία δεν έχουν συμπεριληφθεί γιατί δεν υπάρχει χώρος. Αυτό είναι ο κανόνας του Κοινοβουλίου, να μην το λησμονούμε οι κανονισμοί του Κοινοβουλίου μας έχουν επιβάλει να δουλεύουμε έτσι. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, είναι σημαντικό να μιλήσουμε για αυτές, γιατί έχουμε αρμοδιότητα στον τομέα αυτό. Η Επιτροπή μας και ιδιαίτερα όσο αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπάρχει και η οδηγία για τα ενυπόθηκα δάνεια. Και αυτή είναι μια χρηματοπιστωτική υπηρεσία. Είναι λοιπόν μια αρμοδιότητα για την οποία πρέπει να μιλήσουμε. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι ορθώς ε, γίνεται λόγος για αυτά τα προϊόντα, για αυτές τις υπηρεσίες. Πάρα πολλοί καταναλωτές δεν ε, κατανοούν γιατί, πώς είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για προστασία του καταναλωτού χωρίς να γίνεται λόγος για προστασία των τροφίμων, παραδείγματο χάρη. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που πρέπει να υποθούν. Ωστόσο, εγώ για άλλο λόγο ε, έχω ζητήσει το λόγο. Ε, υπάρχει η επικαιροποίηση και η εκτέλεση. Είναι θεμελιώδη ζητήματα αυτά. Πρέπει να αντιμετωπισθούν. Ξέρω ότι άλλοι δεν έχουν την ίδια άποψη. Ο κύριος Σβάμπ έχει επιφυλάξεις. Ε, αλλά με τις επιφυλάξεις δεν καταφέρνουμε και πολλά. Πρέπει να, έχουμε, να είμαστε θετικοί. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να μπορεί να συναποφασίζει. Ε, δεν έχουμε κατά νου τις συλλογικές αγωγές όπως αυτές εφαρμόζονται στις Ηνωμένε Πολιτείες. Σίγουρα δεν μπορεί να λειτουργήσει ο θεσμός αυτός έτσι εδώ στην Ευρώπη. Δεν το αντέχει και η τσέπη των καταναλωτών. Μόνο η τσέπη των δικηγόρων επωφελείται. Ε, ωστόσο, πρέπει να φροντίσουμε οι καταναλωτές μας ε, να απολαμβάνουν προστασία των δικαιωμάτων τους στην εσωτερική αγορά και πρέπει να θεσπίσουμε και να λειτουργήσουμε τους σωστούς νομικούς θεσμούς και διαδικασίες. Υπάρχουν, ε, υπάρχει εναλλακτική επίλυση διαφορών. να το προωθήσουμε και αυτό. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που δεν αρκούν αυτές οι μέθοδοι αυτός ο τύπος εναλλακτικής διευθέτησης δεν αρκεί σε πολλές περιπτώσεις και υπάρχει ανάγκη να υπάρξουν άλλοι μηχανισμοί και άλλες μορφές προσφυγής στο δικαστήριο. Εγώ προτιμώ τους εναλλακτικού τρόπους διευθέτησης, αλλά όταν αυτοί δεν ευδοκιμούν πρέπει να έχουν δικαιώματα οι καταναλωτές και άλλων μορφών. Θα ήθελα λοιπόν να τύχει μεγαλύτερη επεξεργασία το θέμα αυτό στην έκθεση, αν συμφωνεί και ο εισηγητή. Μάλιστα σήμερα έλαβα ε, την προσφυγή ενός πολίτη, ενός Γερμανού πολίτη που ζει στην Γαλλία και που, έχει, παρήγγειλε κάτι μέσω της ιστοσελίδας Amazon και είδε ότι στην ιστοσελίδα Amazon, στην γερμανόφωνη σελίδα, ε, προσέφερε προϊόντα πολύ καλύτερα και πολύ πιο βολικά από ότι η γαλλική σελίδα. Και έτσι έκανε την παραγγελία του στη γερμανόφωνη σελίδα της Amazon.com. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να παρέμβουμε εδώ. Δεν είναι δυνατόν οι επιχειρήσεις να κρύβονται πίσω από τα εσωτερικά σύνορα εις βάρος των συμφερόντων των καταναλωτών. Και, ως και γι' αυτό επίσης πρέπει να μιλήσουμε, γιατί πρόσφατα πολλοί ε, ε, έχουν παράπονα αυτού του τύπου και ασκούν προσφυγές για αυτόν τον λόγο. Και για παράδειγμα, όταν ε, γίνονται παραγγελίες μέσω δικτυακών τόπων και η παράδοση δεν γίνεται με τον ε, πρέποντα τρόπο. Ε, θυμάμαι, για παράδειγμα, στη Γερμανία ένα συγκεκριμένο προϊόν κόστιζε 200 ευρώ λιγότερο από ό,τι στη Γαλλία. Ε, και εγώ λοιπόν το ίδιο έκανα. Το παρήγγελα στη Γερμανία, το πήρε η μητέρα μου και μου το έστειλε στην Γαλλία. Ε, δεν πρέπει να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην εσωτερική αγορά όμως. Κάτι άλλο που το θέλω ενισχυμένο στο θεματολόγιο για τους καταναλωτές ε, και συγκεκριμένα η εφαρμογή του δικαίου που υιοθετούμε. Διάβαζα στις εφημερίδες τις προάλλες ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα έκανε κάποιους ελέγχους σε δικτυακούς τόπους για να διαπιστώσει αν τηρούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία, συγκεκριμένα δικτυακούς τόπους που προσφέρουν δωρεάν παιχνίδια. Και διαπίστωσε η Επιτροπή ότι υπάρχουν περίπου, υπάρχει περίπου ένα 50% δικτυακών τόπων που απευθύνονται σε άτομα κάτω των 15 ετών που δεν πληρούν τους κανόνες μας. Στην πραγματικότητα πρόκειται για παγίδες. Οι νέοι θεωρούν ότι κάποιο παιχνίδι είναι δωρεάν, το κατεβάζουν από το διαδίκτυο και στη συνέχεια πρέπει να πληρώσουν δαπάνες και φυσικά οι γονείς τους πρέπει να τις καλύψουν. Ε, νομίζω πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας και ασφαλώς Πρέπει ε, κάτι να συμφωνήσουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για να ε, κάνουν κάτι τα κράτη-μέλη, να ενισχύσουν τους ελέγχους τους. Και γι' αυτό πρέπει να γίνει λόγος, πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω πολύ καλά τους περιορισμούς που έχουμε, που έχουν οι εισηγητές σε όλη αυτή την σύνταξη. Όλοι μας οι σκιώδεις εισηγητές έχουμε ρόλο να προσθέσουμε ορισμένα σημεία για να εστιαστούμε σε αυτό που απαιτεί το θεματολόγιο των ε, προστασίας των καταναλωτών. Έχουμε κάνει αρκετή εργασία ε, και είναι ε, σημαντικό να είμαστε θεματοφύλακες των συμφερόντων των καταναλωτών. Ίσως άλλοι άλλη να μην συμφωνούν σχετικά με την άποψη αυτή με συγχωρείτε που δουλέψαμε αποτελεσματικά ε, και τελειώσαμε πιο νωρίς ε, τα προηγούμενα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Ε, σας καλωσορίζω εδώ και θα θέλαμε να έχουμε τα σχόλια σας, τα σχόλια της Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα είμαι εδώ από την Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης από την Κομισιόν ε, διότι το θεματολόγιο ε, της, ε, της, για την κατανάλωση και τους καταναλωτές ανήκει επίσης και στην Επίτροπο Ρέντινγκ. Θέλουμε σε ένα έγγραφο να έχουμε όλη την εργασία της Κομισιόν σε σχέση με τους καταναλωτές. Δεν είναι μόνο λοιπόν η Γενική Διεύθυνση για τους καταναλωτές έχουμε και άλλες γενικές διευθύνσεις, δικαιοσύνη, DigiMove, για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών. Αυτή η ολιστική άποψη ανταποκρίνεται σε έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχουμε μια σφαιρική προοπτική σχετικά με την πολιτική που σχετίζεται με τους καταναλωτές αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτή η έκθεση, το θεματολόγιο πρέπει να το δούμε σε δύο επίπεδα. Πάρα πολλά στοιχεία που έχουμε περιλάβει ισχύουν ε, μέχρι το 2020, τον ορίζοντα 2020, αλλά για συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες μπορούμε μόνο να αναγγείλουμε προτάσεις και πρωτοβουλίες από το σώμα των επιτρόπων που υπάρχει τώρα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν το, και τον ορίζοντα αυτό που είναι το τέλος του 2014. Ε, ε, χαιρόμεθα που ο εισηγητής συμφωνεί με την ασφάλεια, την ενημέρωση, την κατάρτιση, επίσης επιβολή και διόρθωση και προσφυγή με αυτούς τους στόχους και τις προτεραιότητες. Βεβαίως ε, δίνεται μεγάλη έμφαση στην επιβολή ε, του νόμου, στην εφαρμογή, διότι του χρόνου θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με την εφαρμογή και την επιβολή και τα δύο παραδείγματα που έδωσε η κυρία Γκέπχαρντ την ε, διαφοροποίηση των τιμών από την ίδια εταιρεία σε διαφορετικές χώρες, σε διαφορετικές εθνικές αγορές είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει πρόσφατα με, ε, τους, ε, με εθνικά υπουργεία ε, και επίσης τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΚ, διότι έχουμε το άρθρο 20 της Οδηγίας περί υπηρεσιών που απαγορεύει τις διακρίσεις στην παροχή υπηρεσιών χωρίς λόγο αντικειμενικό. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και άλλα παραδείγματα που η DG Market έχει ανακαλύψει, αν θέλετε βρίσκεστε στην Αυστρία και θέλετε μια κρουαζιέρα, την πληρώνετε πολύ πιο ακριβά από την Αυστρία από ό,τι από την Γερμανία. Ε, και αν ε, είστε στα βουνά της Ιταλίας ε, θέλετε και θέλετε εκένωση, πληρώνετε πολύ περισσότερα αν είστε Γερμανός υπήκος. Έχουμε λοιπόν αυτές τις διαφορές στις τιμές των υπηρεσιών. Ασχολούμε αυτό, αυτό το θέμα στα πλαίσια της εφαρμογής της οδηγίας περί υπηρεσιών. Σχετικά με την επιβολή ε, θέλουμε να τονίσουμε το θέμα αυτό θα είναι το θέμα της ε, Συνόδου Κορυφής για τους καταναλωτές του χρόνου και στο τέλος του χρόνου θα έχουμε μια στρατηγική για την επιβολή και εφαρμογή των δικαιωμάτων των καταναλωτών και κάτι που θέλουμε να εξετάσουμε είναι πώς μπορούμε καλύτερα να αντιμετωπίσουμε αυτές τις παραβιάσεις που υπάρχουν σε όλη την κοινότητα. Έχουμε τα SWIPS βεβαίως και σχετικά με τα παιχνίδια που μπορεί κανείς να κατεβάσει από το διαδίκτυο. Και πάρα πολύ συχνά έχουμε τη διαφορετική εφαρμογή. Δεν είναι διασυνοριακή εφαρμογή, δεν είναι μια εταιρεία σε μια χώρα Α που ασχολείται με καταναλωτές στην χώρα Β. Είναι η ίδια εταιρεία που είναι εγκατεστημένη σε πάρα πολλές χώρες ε, και ασχολείται με αυτές τις εσωτερικές αγορές των χωρών και έχει τεχνικές αθέμητες ή απατηλές πρακτικές για τις πωλήσει. Εκεί μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για να συντονίσουμε ε, και να μοιραστούμε τις βέλτιστες ε, πρακτικές σχετικά με την ανόρθωση, την συλλογική, την... είναι μέσα στο πρόγραμμα της Κομισιόν και συζητούμε την μορφή που πρέπει να πάρει ε, με τους συναδέλφους ε, της ε, DG Justice και της DG Competition. Δεν ξέρω εάν θέλει κάτι να προσθέσει ο συνάδελφος από την DG Justice. Ευχαριστώ τους εισηγητές και τους κοιόδης και περιμένουμε την εισήγηση αυτή. Θα δώσω τον λόγο στην Βερόνικα Φρέντι που θέλει κάτι να προσθέσει. Νομίζω, όχι. Όχι, όχι, δεν υπάρχουν πολλά ε, να προσθεθούν σε αυτά που μόλις τώρα λέχθηκαν. Υπάρχουν μερικές ιδέες που χρειάζονται περαιτέρω συζήτηση. Ε, οι αντιπρόεδροι ε, έχουν ε, την ε, πρωτοβουλία Women on Board και λάβαμε υπόψη το γεγονός ότι ο εισηγητής θέλει ίσως μερικούς καταναλωτές στα συμβούλια των εταιριών. Αυτό χρειάζεται κάποια συζήτηση το θέμα. Αυτό είναι κάτι το πολύ τολμηρό θα έλεγα. Έχουμε πλήρη υποστήριξη για ό,τι είπε η κυρία Μάινορ και η DG Anchor ε, χρειάζεται ε, να ενισχύσουμε εδώ το θέμα της επιβολής ε, το τμήμα του κεκτημένου που δεν εφαρμόζεται. Θα πρέπει να ξανασκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι εθνικές δυνάμεις, κυρίως λαμβάνοντα υπόψη τις εξελίξεις στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ και τις δυο σας. Νομίζω ότι μας δώσατε μερικές ακόμη ιδέες που μπορούμε να σκεφτούμε και να ενισχύσουμε τα όσα είπε ε, η κυρία Γκέπχαρτ ε, για τα θέματα αυτά των SWIPs ε, διασυνοριακά και επίσης για διαπιστώσεις καταναλωτών. Θα δίνω τώρα τον λόγο στον εισηγητή που θα συνοψίσει και θα σχολιάσει ορισμένα από τα σημεία και να μιλήσει για το χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα στάδια αυτής της εισήγησης. Έχετε το λόγο κύριε εισηγητά. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Μια γενική παρατήρηση πρώτα απ' όλα παρακαλώ. Μιλάτε για τον ολιστικό χαρακτήρα του θεματολογίου για τους καταναλωτές. Όντως είναι κεντρική σημασίας Δίχως άλλο, αυτό σημαίνει ότι βλέπουμε τον καταναλωτή σαν τον πυρήνα του οικονομικού συστήματος και σαν ένα όλο, σαν ένα σύνολο. Τον καταναλωτή πολίτη. Ωραία. Και είναι πολύ σωστό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου που συζητάμε. Δεύτερη γενική παρατήρηση. Ο τρόπος που έχει γίνει η διατύπωση στην πρότασή μου και το εύρος της. Τώρα που έχω ακούσει τους σκιώδεις εισηγητές, νομίζω ότι θα είναι εύκολο να καταλήξουμε σε συμφωνίες. Το να υπάρχει καλύτερη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων μερών και μια διατύπωση ε, πιο κατάλληλη για όλους είναι κάτι που πιστεύω ότι θα επιτευχθεί εύκολα. Θα φροντίσω να έχουμε μια συνάντηση με τους σκιώδεις εισηγητές τις επόμενες ημέρες. Να τηρήσουμε φυσικά βέβαια και το ημερολογιακό έτος, έτσι. Και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Μια άλλη γενική παρατήρηση που έχω να κάνω είναι το ότι όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς υπάρχει περιορισμός στην έκταση της πρότασης όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Δεν μπορούσα να τα συμπεριλάβω όλα, ακόμα και αν συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπατε εσείς, εγώ δεν μπορούσα να τα συμπεριλάβω λόγω περιορισμού ε, έκτασης της πρότασης που μου επιβάλλεται. Με τροπολογίες, εσείς είτε κι εγώ μπορούμε να συμπληρώσουμε την πρότασή μου προς την κατεύθυνση που επιθυμείτε, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Αυτές είναι οι γενικές μου παρατηρήσεις. Τώρα, πιο συγκεκριμένα για τα σχόλια που κάνατε. Έχω να πω τα Μου ζητήσατε να λάβω υπόψη μου ότι τη σήμερον ημέρα δεν θα έπρεπε να επιφορτίζουμε με επιπλέον κόστος τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνοι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραβιάζονται τα δικαιώματα των καταναλωτών από την άλλη. Άρα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια καλή συμφωνία. Για μένα προτεραιότητα Στη σημερινή οικονομική κατάσταση που βρισκόμαστε, για μένα λοιπόν προτεραιότητα είναι τα δικαιώματα των καταναλωτών. Δεν νομίζω, από την άλλη, ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να κάνουμε προτάσεις στο θεματολόγιο για τους καταναλωτές, αν δεν λάβουμε υπόψη μας την πραγματικότητα που ζει σήμερα ο καταναλωτής, αλλά και τις προοπτικές που έχει για το μέλλον. Εμείς πρέπει να υπογραμμίζουμε τις απαιτήσεις και τις προτάσεις που υποβάλλουν οι καταναλωτές και μας στέλνουν αυτή την περίοδο. Για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, το είπατε και συμφωνώ, ότι δεν μπορούμε να το αποφύγουμε πρώτα απ' όλα. Οπότε ας συμφωνήσουμε τι πρόταση θα κάνουμε. Δίχως άλλο όμως, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα και απασχολεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Τώρα διάφοροι σκιώδεις εισηγητές είπατε ότι κάποια σημεία στην έκθεσή μου έχουν να κάνουν με την ισπανική πραγματικότητα. Μπορεί. Η οικονομική κατάσταση βέβαια δεν είναι ίδια στις 27 μας χώρες Υπάρχει όμως ένας ελάχιστος κοινό παρονομαστής, που είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι οικονομικοί, δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές σήμερα. Δεν νομίζω ότι επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ μας, δεν πρέπει να επιμείνουμε στις απαιτήσει και στις επιθυμίες των καταναλωτών που προέρχονται από ολόκληρη την Ευρώπη και που είναι κοινέ. Τώρα από τις προτάσεις μου. Η πρότασή μου αριθμός 3. Τι είπατε για αυτήν. Εδώ νομίζω ότι πρέπει πράγματι τις επόμενες μέρες να διευκρινίσουμε τι είναι το Μητρό Ευρωπαϊκών Ενώσεων. θα πρέπει να είναι κάτι όπως ε, αναφέρεται στην οδηγία 22 του 2009 που μιλάει για την εναρμόνιση των ελάχιστων δικαιωμάτων των ε, Ευρωπαϊκών Ενώσεων Καταναλωτών. Ότι δηλαδή πρέπει να έχουμε διαβούλευση μαζί τους και να ακούμε την απόψή τους. Σημείο 6 που αναφέρατε επίσης. για την εχναλυσιμότητα. Θέλετε τον όρο αυτό. Καλώς. Σημείο 8 και 10. Εδώ αναφέρομαι στην σημερινή πραγματικότητα και στην ανησυχία των καταναλωτών όσον αφορά τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αλλά αναφέρομαι επίσης και στην κατοικία τους. Εδώ είμαι ανοιχτό, εφόσον θέλετε, να προσπαθήσουμε να βρούμε μια διατύπωση που να είναι περισσότερο κατανοητή. Σημείο 15. Σίγουρα είναι τολμηρό. Το να μιλάμε για 20% εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να τολμάει. Στο κάτω-κάτω αυτά είναι πράγματα τα οποία ζητάει ο κόσμος η πλειοψηφία των καταναλωτών, άρα πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτά που θέλουν. Τώρα για τις συλλογικές ε, προσφυγές. Το θεματολόγιο για τους καταναλωτές πρέπει να το συμπεριλαμβάνει αυτό για να βελτιωθούν οι εγγύησει για τις συλλογικές προσφυγές των καταναλωτών να διευκολύνεται δηλαδή η πρόσβαση των καταναλωτών στους μηχανισμούς αυτούς, να είναι αποτελεσματικές αυτές οι μέθοδοι, ε, να περιορίζεται ο χρόνος, να μην υπάρχει καθυστέρηση δηλαδή. Αλλά και εδώ μεταξύ μας θα προσπαθήσουμε να βρούμε την καλύτερη δυνατόν διατύπωση για να βελτιωθεί αυτό το σημείο. Ίσως θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τη δυνατότητα των μηχανισμών διαιτησίας που θα υιοθετηθούν να ε, μπορεί να υπάρξει στα πλαίσια αυτά η προσφυγή. Τώρα κάτι άλλο που ανέφεραν διάφοροι σκιώδεις εισηγητές είναι ότι υπάρχουν καινοτομίε μέσα στην ε, εκθεσή μου, δηλαδή ότι μιλάω για την υγεία ή για άλλα θέματα που ίσως δεν αφορούν άμεσα τα δικαιώματα καταναλωτών. Ναι, αλλά από την άλλη, αυτά απασχολούν τους καταναλωτές και γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις. Λίγο πολύ, αυτά δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι, αλλά νομίζω ότι τα πιο σημαντικά τα απάντησα. Πάντως επιμένω ότι είμαι στη διάθεσή σας για να πετύχουμε συμφωνίες μεταξύ μας ίσως να συναντηθούμε σύντομα οι σκιώδες εισηγητές και να προσπαθήσουμε με τροπολογίες να βρούμε το καλύτερο τρόπο για να βελτιωθεί τελικά η έκθεση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, ευχαρίστω να ακούσω και τις προτάσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Είμαι στη διάθεσή σας και γι' αυτό και πάλι με στόχο να πετύχουμε την καλύτερη πρόταση για το ευρωπαϊκό θεματολόγιο του τους Μου είπατε να μιλήσω για το χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 10 Ιανουαρίου. Εντάξει, πρέπει να βιαστούμε. Δεν έχουμε μεγάλο περιθώριο για τον κοινοβουλευτικό διάλογο, αλλά αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Και ας προσπαθήσουμε σε αυτό το διάστημα να πετύχουμε όσο γίνεται πιο ευρεία συνένεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η ευκαιρία για συζήτηση. Κουβέντιαζα εδώ ε, για την δυνατότητα να αναβάλουμε λίγο την ε, προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Νομίζω ότι οι σκιώδεις εισηγητές θα χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να υποβάλουν τροπολογίες που να συμπεριλάβουν όλα αυτά τα οποία είπαμε. Νομίζω ότι θα είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Η σύστασή μου είναι λοιπόν να συζητήσετε μεταξύ σας και αύριο το απόγευμα στη συνεδρίαση των ε, συντονιστών να το δούμε. Να έχουμε ας πούμε ως προθεσμία την 25η Ιανουαρίου. Δεν νομίζω ότι πρόκειται να συναντηθούμε πριν το τέλος αυτής των εργασιών του Κοινοβουλίου την Τετάρτη. Κύριε Γκαρσές Ραμόν, αν συμφωνείτε με αυτό, θα προσπαθήσουμε να σας βρούμε λίγο περισσότερο χρόνο. Μάλλον θα συμφωνήσετε βέβαια. Θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι είναι καλή ιδέα. Ναι, ναι, ασφαλώς βρίσκω ότι είναι πολύ καλή ιδέα και τη στηρίζω απόλυτα. Εντάξει, θα το συζητήσουμε και αύριο με τους, συντονισμέ, με τους συντονιστές θα δούμε πού θα μπορέσουμε να το στριμώξουμε για να μπορέσουμε να σας δώσουμε χρόνο να συμπεριλάβετε τις ιδέες τόσο της κυρίας Μάιναρ όσο και της κυρίας Μανφρέντι που είναι πάρα πολύ χρήσιμες και ευπρόσδεκτες και τουλάχιστον να αξίζει τον κόπο η τρεχάλα τους μέχρι εδώ. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ γι' αυτό. Έχουμε προχωρήσει στο χρόνο, αλλά για να ελέγξω αν έχουμε εδώ όλους τους σχετικούς με τη συζήτηση για τα προσωπικά δεδομένα. Για να δω ποιοι είναι εδώ. Η κυρία Ρούλη ήταν πριν εδώ, τώρα δεν είμαι... Ο κύριος Ροσφόρ θα μιλήσει στη θέση του κύριου Λούφιγκα. Εδώ, εγώ είμαι ένας από τους σκιώδεις εισηγητές της ομάδας μου. Και έχουμε και την κυρία Βιντονσέ μαζί μας. Κυρία Βασιλείου, αν δεν κάνω λάθος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σπεύσατε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε εδώ μαζί μας παρατάθηκε πολύ η συνδιάσκεψη των Προέδρων, ήταν μακρά η ημέρα σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, όλοι εδώ είναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θα δώσω τον ε, λόγο στην κυρία Κόμη για να παρουσιάσει τις συμβιβαστικές της προτάσεις και να μας πει και ό,τι άλλο θέλει. Στη συνέχεια οι σκιώδεις εισηγητές ε, θα λάβουν τον λόγο και μετά θα έχουμε χρόνο για ερωτήσεις και απαντήσεις. Πρώτα λοιπόν ο λόγος στη Λάρα Κόμη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για την συνεργασία σας μέχρι στιγμής. Είμαι πολύ ευτυχής με τον τρόπο που εργαστήκαμε. Φτάσαμε σε συμφωνία πάνω σε πολύ σημαντικά θέματα. Το θέμα πάνω στο οποίο εργαζόμαστε αποδείχτηκε ανοιχτό στη συνεργασία και στη συζήτηση. Και έτσι πραγματικά εργαστήκαμε με, μεγάλο, με μεγάλη ζέση και ευρηματικότητα. Όπως ξέρετε, μιλούμε για την προστασία των καταναλωτών χωρίς να χάνουμε από μπροστά μας τη συνοχή της αγοράς η συζήτηση επίσης πολύ λίγο προσέκρουσε σε ιδεολογικά προσκόμματα και γι' αυτό έχουμε προχωρήσει πολύ ικανοποιητικά. Ένα ευαίσθητο θέμα που έχει να κάνει με την προσωπική ευαισθησία, με την εμπειρία του καθενός μας, η ιδέα της προστασίας σε εθνική βάση, σε πολιτική βάση. Απευθύνω έκκληση σε όλους τους συναδέλφους να υιοθετήσουμε μέτρα που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και να βάλουμε κατά μέρο τις προσωπικές μας εμπειρίες που θέτουν σε κίνδυνο τον κανονισμό αυτόν. Εμείς θέλουμε να προάγουμε μια εσωτερική αγορά. Υπάρχει αυτή η μεθοδολογική αρχή, την οποία ήθελα να παρουσιάσω εν είδη εισαγωγής, γιατί πραγματικά συναντήσαμε πάρα πολλά εμπόδια, εμπόδια εθνικής και πολιτισμικής υφής. Θα ήθελα ε, να αναδυθούν οι διαφορές που μέχρι στιγμής εμπόδισαν τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Εάν συμφωνείτε θα ξεκινήσω από την κατάρτιση προφίλ. Θα ήθελα η Επιτροπή να παρέμβει στη συνέχεια και να διευκρινίσει τι θέλει να ρυθμίσει όταν συνέταξε το άρθρο 20. Γιατί φοβάμαι ότι υπάρχει ένα ουσιώδες θέμα και εξηγούμε. Δεν θέλω να φανώ ότι εκπροσωπώ μια αλήθεια που δεν υπάρχει. Μακριά από μένα αυτή η ευθύνη. Δεν θέλω να πω ότι οι άλλοι συνάδελφοι έχουν λιγότερο δικαίωμα να θελήσουν να ρυθμίσουν πτυχές άλλες από αυτές που θέλω εγώ. Θέλω να πάω πέρα από τις ιδεολογικές διαφορές και να επιχειρηματολογήσουμε μαζί για να καλύψουμε όλα τα θέματα που δεν υπόκεινται σε πεδίο αρμοδιοτήτων άλλων επιτροπών και υπηρεσιών. Θα κάνω συγκεκριμένα παραδείγματα, θα φέρω συγκεκριμένα παραδείγματα για να αναδείξω τις δικές μου δυσκολίες και τις δυσκολίες που συνάντησαν οι άλλοι. Για την κατάρτιση προφίλ, τι εννοούμε, την κατηγοριοποίηση που γίνεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες για τη διαχείριση κινδύνου, για τη διαπίστωση κινδύνου. Δεν μπορώ να φανταστώ ποιοι κίνδυνοι εκπορεύονται από αυτό το σύστημα όταν υπάρχει και το opt-out. Άλλο παράδειγμα. Αν εννοούμε την κατηγοριοποίηση από την συμπεριφορά marketing, δύο πράγματα να πούμε. Προτιμώ όταν γίνεται διαφήμιση για τσάντες ή για παπούτσια ή για φαγητά ε, ε, πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Δεν μπορούμε να ρυθμίζουμε μόνο τα εμπορεύματα που μας αρέσουν και όχι εκείνα που δεν μας αρέσουν. Υπάρχει δυνατότητα αντίρρησης στην επεξεργασία δεδομένων. Άρθρο 19. Υπάρχουν και τα δεδομένα του άρθρου 16. Υπάρχει μια αναντιστοιχία μεταξύ των δύο. Άλλο παράδειγμα, μπορώ να φέρω κι άλλα βέβαια. Με συγχωρείτε πάρα πολύ που γίνομαι τόσο συγκεκριμένη, αλλά θέλω να επικαλούμε την πραγματικότητα για να δείξω ποιες είναι οι δυσκολίες. Εάν σε μία μηχανή έρευνη, σε ένα ψαχτήρι ιταλικό, ε, ψάχνω στην Ιταλία μόνο, εξοικονομώ χρόνο και κόπο, ε, βάζοντας και άλλες παραμέτρους έρευνας ανάλογα με τα κριτήριά μου και τις προτιμήσεις μου. Θέλω να ξεκαθαρίσω μαζί σας και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τους κοιόδης εισηγητές ποια είναι η πραγματική αξία της κατάρτισης προφίλ άλλο στοιχείο, όπου υπάρχουν ιδεολογικές αντιρρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. παρόλες τις κανόνες, κανονισμούς, οδηγίες, συστάσεις, πάντοτε υπάρχει η δυσκολία να βρούμε τον σωστό τρόπο βοήθειας και στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γι' αυτό εγώ προσπάθησα να ακυρώσω εκείνους τους κανόνες που έθεταν κάποιο κατόφλι για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, αλλά συνδέεται κυρίως με άλλους παράγοντες. Και γι' αυτό Χρειάζομαι λίγο περισσότερο χρόνο για να βρω παραμέτρους και να τους προτείνω αργότερα. Μερικές φορές είναι πολύ μηχανιστικοί οι παράμετροι εφαρμογής. Είναι ανεφάρμοστη, τι. Πάνω σε αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να λάβει το λόγο. Στους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες τέτοιες, ρωτώ, θέλουμε πραγματικά και άλλο ένα πρακτικό παράδειγμα. Ε, έχει τις ίδιες υποχρεώσεις ε, και το υπόκειται στο ίδιο κόστος το μαγαζάκι της γωνιάς της γειτονιάς μας και, και μια μεγάλη εταιρεία. Μια εταιρεία που απασχολεί 50 με 60 εργαζομένους είναι μια μεγάλη επιχείρηση, δεν είναι μικρομεσαία επιχείρηση. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. δεν θέλω να αποσύσω την ευθύνη που ανήκει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, χειροτεχνίες, βιοτεχνικές ε, επιχειρήσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις, ε, ή ακόμα και βιβλιοπόλες. Το άτομο που διαχειρίζεται ε, τα άτομα το άτομο που διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να μάθει να ενεργεί με ορισμένα κριτήρια. Έχω συζητήσει με τον συνάδελφο από την Επιτροπή Ελευθεριών για η προστασία των ανηλίκων είναι σίγουρα στόχος όλων μας η προστασία των ανηλίκων, γιατί είναι μια κατηγορία καταναλωτών πολύ πιο ευαίσθητη. Υπάρχουν όμως αμφιβολίες πρακτικού χαρακτήρα. Όταν ένα εθνικό νομοθέτημα λέει ότι στα 17 έτη μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, μπορεί να παντρευτεί, μπορεί να κάνει παιδιά, αλλά χρειάζεται ειδική μεταχείριση όταν αφορά για, την, για τη διαγραφή προσωπικών στοιχείων, μου φαίνεται ότι αυτό είναι μια αντίφαση. Στα 17 πολλές φορές δίνουμε μεγάλες υπευθυνότητες στους ανηλίκους. Και θα πρέπει ίσως να ζητείτε η συγκατάθεση των γονέων. Δηλαδή για να παντρευτούν δεν χρειάζονται τη συγκατάθεση των γονέων, αλλά για να διαγραφούν τα προσωπικά του στοιχεία χρειάζεται η συγκατάθεση των γονέων ενημέρωση. Το θέμα της ενημέρωσης πρέπει να είναι πολύ... πάνω στο θέμα της ενημέρωσης πρέπει να ενσκύψουμε πολύ. Έχει να κάνει και με την δημοκρατική λειτουργία των θεσμών. Ωστόσο, ήθελα να φέρω σε προσοχή σας όλες αυτές τις προβληματικές. Δεν είναι εθνικά προβλήματα. Είναι προβλήματα που ανακύπτουν στην εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά. Σταματώ εδώ με χαρά θα ακούσω τις ε, θέσεις των συναδέλφων, τους οποίους ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη γόνιμη συνεργασία τους και για την βοήθειά τους. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Mrs. Kami. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κάμι. Ε, κυρία Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Κόμη με συγχωρείτε, η φωνή μου δεν είναι τόσο καλή σήμερα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι είχαμε πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων στο Στρασβουργό σχετικά με τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Αλλά όπως είπα, κατά τη διάρκεια αυτής της ανταλλαγής απόψεων δεν είχαμε αποφασίσει ε, για τις συμβιβαστικές τροπολογίες στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και έχουμε μερικές αμφιβολίες ακόμα και γενικά θα πρέπει να δούμε πώς, ποια είναι η θέση σας σχετικά με πολλές τροπολογίες που είναι σημαντικές για την ομάδα μας. Για την ώρα είναι δύσκολο για μας να υποστηρίξουμε όλες τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Αυτό που είναι σημαντικό για μας ε, όσον αφορά την συζήτηση για την συνένεση, τη συγκατάθεση, είναι ε, να αφήσουμε την δυνατότητα για ρητή συγκατάθεση. Είναι στον συμβιβασμό 1 και 6 αλλά είναι μόνον όταν πρόκειται για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. Επίσης ε, έχουμε μερικά προβλήματα για τον ορισμό ε, των συζητουμένων θεμάτων. Τα, ε, στους δεν περιλάβατε καμιά τροπολογία της σοσιαλιστικής ομάδας. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να εργαστούμε για αυτές. Αναφέρατε το θέμα της ηλικίας. Συμφωνούμε ότι υπάρχουν ορισμένα προβλήματα με τον ε, ορισμό ότι επειδή έχουμε πάρα πολλούς διαφορετικούς ορισμούς σχετικά με τους νέους στην Ευρώπη, αλλά πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε προστασία των παιδιών μέχρι την ηλικία των 18. Είμαστε, ε, πολύ, ε, είμαστε μάλλον υπέρ του αρχικού κειμένου της Επιτροπής που καλύπτει το θέμα αυτό καλύτερα από τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Σχετικά με το profiling, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ορισμένα προβλήματα με την πλήρη κατανόηση του θέματος. Ε, μερικοί, συμβιβασμοί αναφέρονται ε, στην διαγραφή της δυνατότητας των καταναλώδων να έχουν opting out από μέτρα profiling ε, για να απαγορευθούν ορισμένες διακρίσεις. Αυτό δεν είναι καλό για μας, αλλιώς θα αρχίσουμε να συζητούμε πότε είναι δίκαιο, πότε είναι διάκριση κλπ. Νομίζουμε ότι είναι πολύ ευρύ το θέμα, γι' αυτό είναι καλύτερα να δώσουμε στους καταναλωτές μια επιλογή, μια δυνατότητα επιλογή, ένα opting out. Ε, μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε αυτό και συζητήσαμε επίσης τις παραβιάσεις δεδομένων και αν θα υπάρχει ένας χρονικός περιορισμός ή όχι. Και επίσης πιστεύουμε ότι θα πρέπει να βρούμε εδώ έναν περιορισμό χρόνου συγκεκριμένο. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να εργαστούμε για ορισμένα από τα προβλήματα για να προχωρήσουμε. Επίσης, κατάλαβα ότι δεν μπορείτε να υποστηρίξετε τις τροπολογίες που είχαμε σε σχέση με τις ε, συλλογικές ε, συμφωνίες και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ομάδα μας, ούτε ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε υπέρ του συνόλου της εισήγησης. Απλώς θέλω λοιπόν να πω, είχαμε πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων στο Στρασβούργο και ε, νομίζω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μερικά από αυτά τα θέματα αν έχουμε ε, μια ε, πραγματική συνεδρίαση, συνάντηση και όχι ανταλλαγή απόψεων ε, ηλεκτρονικά. Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε, αλλά θέλουμε κάποια κίνηση προς την πλευρά μας για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε το κείμενο. Νομίζω ότι αυτό είναι εφικτό και μπορούμε να βρούμε καλούς συμβιβασμούς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, βεβαίω έχουμε την ψηφοφορία στις 24 Ιανουαρίου, έχουμε χρόνο για περαιτέρω συζήτηση. Είναι καλό που έχουμε αυτούς του συμβιβασμούς ε, που εκφράστηκαν αρκετά νωρί για να μπορούν να αποφανθούν όλες οι ομάδες. Έχουμε βεβαίω ε, μερικέ λεπτομερείς, θέματα. Τώρα, ο κύριος Ροσφόρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Λοκογκάρτ έπρεπε να είναι εδώ. Εγώ τελευταία στιγμή αναγκάστηκα να τον αντικαταστήσω. Μου διαβίβασε ένα σημείωμα όπου σχετικά με τις συμβιβασμούς έτσι όπως κατέληξαν σήμερα δεν είναι βέβαιος ότι έχει εξετάσει τα πάντα και δεν έχει λάβει θέση για όλα. Ευχαριστεί την εισηγήτρια, την κυρία Κόμη, που προσπάθησε να βρει συμβιβασμούς που βρίσκει λογικούς για θέματα πάρα πολύ σημαντικά, τους μηχανισμούς ε, έγκρισης, το profiling για το οποίο μιλήσαμε, ο κύριος Λεκογκάρτ ε, ε, εγκρίνει και αυτά τις, αυτούς τους συμβασμούς και τις κυρώσεις ε, για τις επιχειρήσεις πολύ καλά επειδή υπάρχουν συμβιβασμοί για την παρότριση επιχειρήσεων να σκεφτούν μέτρα προστασίας ε, των δεδομένων στη φάση συγκρότησης των συλλογών δεδομένων με τους χρήστες και τους καταναλωτές και το γεγονός ότι ενθαρρύνεται ε, μια εισαγωγή μηχανισμών προστασίας αρκετά στερεών για να μπορέσουμε να προαγάγουμε τις διαδικασίες ανομινιμοποίησης των ε, δεδομένων. Ένα αίτημα ε, διαβιβάζω εκ μέρους του κυρίου Λεκογκάρτ στην εισηγήτρια είναι το γεγονός ότι από τη δική του άποψη η πρόληψη των, της απάτης και της οικονομικής εγκληματικότητας του φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερη σημασία τέτοια σημασία, ώστε ε, αυτό περνάει στο άρθρο 6 από τις αιτιολογικές σκέψεις. Να μπει στο άρθρο 6 είναι ένα διακύβευμα ιδιαίτερα σημαντικό για την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Και όπως ε, ελέγχθηκε ήδη τώρα, ε, έχουμε λίγο χρόνο για να οριστικοποιήσουμε όλους τους συμβιβασμούς και ο κύριος Λεκογκάρτ έχει εμπιστοσύνη ότι θα καταλήξουμε σε αποτελέσματα θετικά ε, στις επόμενες συνεδριάσεις που θα λάβουν χώρα στην αρχή του μηνός Ιανουαρίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Άγκστρομ. Ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο, σύντομο με τον προλαλήσαντα ε, νομίζω μια άλλη συνεδρίαση ή ε, εισηγητών θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Σύμφωνο και μαζί σας. Ε, περιορίζω το σχόλιο μου σε αυτό. Ναι, ναι, ενηγματική η συμβολή σας. Καλά, θέλω να πω ότι κάποια μου φαίνονται καλά, κάποια άλλα ίσως πρέπει να τα συζητήσουμε και δεν είμαι 100% σίγουρος για το ότι εννοείται πίσω από αυτά που προτείνεται. Γι' αυτό. Πρόεδρος. Εκ μέρους της δικιάς μου ομάδος. Συμφωνούμε και με τους προλαλήσαντες ότι πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω πάνω σε αυτά. Το σημαντικό πάντως είναι ότι η κυρία Κόμη όντως εντοπίζει τα πιο σημαντικά θέματα, γι' αυτό και τα συζητάμε. Τώρα οι μορφές συνένεσης. Είναι ζωτική σημασία πράγματι. Τη συζήτηση αυτή την έχουμε κάνει και παλιότερα. Με τις μεταρρυθμίσεις για τις οδηγίες όσον αφορά τον ιδιωτικό βίο, με cookies που εμφανίζονται στα κομπιούτερ και πώς θα έπρεπε ο καταναλωτής να ενημερώνεται. Με τέτοιο τρόπο όμως που η αίτηση να γίνεται ρεαλιστικά και τελικά να μην διακόπτει όλη τη διαδικασία συναλλαγής. Ένα πάντως από τα θέματα που τίθενται τώρα είναι ότι οι απαιτήσει για την προστασία του ιδιωτικού βίου φαίνεται να εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο από χώρα σε χώρα. Και εκεί είναι που υπάρχει πρόβλημα νομικής βεβαιότητας. Πρέπει να υπάρχει κάποια συνοχή, γιατί μιλάμε για κανονισμό, δεν μιλάμε για οδηγία. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θα έπρεπε να δούμε. Τις κατευθυντήρες γραμμές δηλαδή για την εφαρμογή το άρθρο 29 για την εφαρμογή όσον αφορά την οδηγία για τα cookies και έτσι να σχηματίσουμε και κάποια συγκεκριμένη εικόνα για το τι είναι πρακτικά εφικτό, ποιες είναι οι προσδοκίες των καταναλωτών που θέλουν να έχουν ενημέρωση, να ελέγχουν τις πληροφορίες κτλ. Αλλά από την άλλη μεριά δεν θέλουν κάθε τρεις και λίγο να βγαίνει κάτι που να του ζητάει ε, στον υπολογιστή να δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Και βέβαια πάντα αυτό είναι ο κίνδυνος, ότι αν αρχίσεις και ζητάς και ξαναζητάς, ε, στο τέλος σε αγνοεί ο καταναλωτής. Οπότε εκεί είναι που καταλαβαίνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προτάσεις της. Πάντως κανείς μας δεν θεωρεί ότι είναι όλα σωστά στην ε, τρέχουσα διατύπωση. Και αυτό ισχύει και για την κατάρτιση προφίλ για το profiling. Εδώ πρέπει να υπάρχουν ρήτρες ασφαλείας. Και με εκπλήσει λίγο το γεγονός ότι βλέπω κάποια μέτρα στην πρόταση της Επιτροπής που το συνδέουν το θέμα με τα θεμητά συμφέροντα, το τι ισχύει στις χώρες μέλη. Αλλά εδώ φοβάμαι ότι καταλήγουμε σε έλλειψη συνοχής με αυτό. Και όπως σας είπα, θέλουμε αποτελεσματικότητα, άρα πρέπει να υπάρχει συνοχή. Τέλος, για την αναλογικότητα. Κάναμε κάποιες προτάσεις, η κυρία δηλαδή, που πάνε προς την σωστή κατεύθυνση, νομίζω, για τις παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων Έχουμε κάποια πράγματα στην οδηγία για τον ιδιωτικό βίο που τα έχουμε περάσει και εδώ. Νομίζω ότι υπάρχει μια καλή ισορροπία. Το πρώτο στοιχείο πάντως της ε, εφαρμογής ε, θα πρέπει να είναι οι αποδείξεις που δεν έχουμε πάντα Όταν ε, συζητούσαμε για την οδηγία για τον ιδιωτικό βίο, το θέμα ήταν η κοινοποίηση. Πώς δηλαδή κοινοποιούνται οι παραβιάσεις της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Έρχονται από τους καταναλωτές. Σίγουρα υπάρχουν πολλές κοινοποίησεις που έρχονται από τους καταναλωτές, αλλά δεν είναι το μόνο. Υπάρχουν μερικά σοβαρά θέματα για τα οποία βέβαια προχωράνε σε κάποια ενέργεια. Αλλά και τα άλλα, πάντα για την αναλογικότητα, υπάρχει και το θέμα των κυρώσεων. Αυτό που προτείνει η κυρία Κόμη πιστεύω ότι πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Και εμεί υποβάλαμε διάφορες τροπολογίες, αλλά πάση περιπτώσει εγώ πιστεύω πως το βασικό εδώ είναι τι επίπτωση έχει η παραβίαση κάθε φορά ανεξάρτητα από το μέγεθος της οργάνωσης που εμπλέκεται, της ε, επιχείρησης που εμπλέκεται. Γιατί ακόμα και μια μικρή επιχείρηση μπορεί κάλλιστα να χειραγωγήσει δεδομένα, ε, να προχωρήσει δηλαδή σε παραβίαση προσωπικών δεδομένων για να υποφεληθεί από αυτό. Δεν είναι επειδή είναι μικρή που δεν ε, θα έχει την πονηριά να το κάνει από την άλλη μεριά μια μεγάλη επιχείρηση. Κατά λάθο. Δεν συμμορφωθεί με κάποιο κομμάτι της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εκεί πρέπει να ληφθεί υπόψη η αναλογικότητα, τη ζημιάς δηλαδή που έχει γίνει. Μιλάτε για πρόστιμα σύμφωνα με τον τζίρο μας, σας λέω, μπορεί να είναι μια μικρή επιχείρηση η οποία μπορεί να κάνει κάτι που έχει ελάχιστε επιπτώσει, αλλά μπορεί να κάνει και κάτι που έχει τεράστιε επιπτώσει. Τι κάνουμε τότε. Πώς σεβόμαστε την αρχή της αναλογικότητας και των προστίμων που επιβάλλονται. Εμείς θέλουμε ε, ο καθένας που μπορεί να έχει στη διάθεσή του προσωπικά δεδομένα να τα μεταχειρίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που λέμε. Άρα πρέπει να βρεθούν οι κατάλληλες διαδικασίες ελέγχου και οι κατάλληλοι επόπτες. Αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Οπότε, σίγουρα υπάρχει κάποια πρόοδος, πάντως σίγουρα η Λάρα Κόμιν διατεθειμένη να συνεργαστεί μαζί μας ε, μέχρι τις 24 Ιανουαρίου, ώστε να έχουμε μια γερή συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων είναι και ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε ότι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα λάβει υπόψη της αυτά που λέμε εμείς. Άλλος κανείς εδώ, παρακαλώ. Έχετε το λόγο εσείς, η Επιτροπή να σχολιάσει. Και μετά η κυρία Κόμη πάλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, εμείς από την πλευρά της Κομισιόν θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε διότι προχωράμε πάρα πολύ ε, γρήγορα. Υπάρχουν κείμενα συμβιβαστικά και είμαστε διαθέσιμοι, είμαστε στη διάθεσή σας. Αναπαιτούνται τεχνικές διευκρινήσεις για την προετοιμασία αυτών των συμβιβαστικών τροπολογιών. Θα προσπαθήσω να επανέλθω σε ορισμένα σημεία χωρίς να μακρηγορήσω. Από γενικής άποψης ε, για την Κομισιόν πρέπει να κρατήσουμε το επίπεδο της 9546 της οδηγίας της ε, υφιστάμενης να κρατήσουμε το επίπεδο προστασίας της υφιστάμενης οδηγίας και είμαστε κάπως επιφυλακτικοί για ό,τι θα συνεπαγόταν μείωση του επίπεδου προστασίας. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που ήθελα να επισημάνω. Δεύτερο, άκουσα για την, την έννοια α, ε, της ρητής συγκατάθεσης. Ακούω κάτι, κάτι που σφυράει. Υπάρχει ένας περίεργος θόρυβος, ενοχλητικός. Δεν τον ακούτε. Η έννοια λοιπόν της συγκατάθεσης που όπως είπαμε η συγκατάθεση είναι από τα θεμέλια της νομιμότητας που επιτρέπει την επεξεργασία των δεδομένων. Αυτό που ήθελε η Κομισιό να κάνει με αυτή την πρόταση είναι να διευκρινίσει ότι αν η συγκατάσταση είναι αναγκαία για κάποια επεξεργασία θα πρέπει να είναι καλή συγκατάθεση. Ε, ναι, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, δεν ακούω πια τα σφύριγματα. Όταν λοιπόν έχουμε συγκατάθεση πρέπει να είναι μια καλή συγκατάθεση και γι' αυτό είχαμε εισαγάγει την έννοια της ρητής συγκατάθεσης. Τώρα και αυτό αναφέρεται σε αιτιολογικές σκέψεις του κειμένου, συμφωνούμε με τα σχόλια σύμφωνα με τα οποία η, ε, ο, δεν πρέπει να είναι ε, να μην ε, να καταστρέφει αυτή η συγκατάθεση της διαδικασίας επεξεργασίας και μια συγκατάθεση θα πρέπει να καλύπτει πολλές δραστηριότητες που έχουν τον ίδιο στόχο. Πράγμα που αναφέρεται σαφώς στις αιτιολογικές σκέψεις είναι ότι πρόκειται για μια συγκατάθεση που μπορεί να εκφραστεί ε, με εστίαση σε ένα κυβότιο ε, διαδικτύου ή με άλλο τρόπο που εκφράζει τη βούληση, ούτω ώστε να καταλάβουμε ότι ένα άτομο δέχεται την επεξεργασία δεδομένων σχετικά με τις διάφορες παρατηρήσεις ε, για την ισορροπία των συμφερόντων και τις βάσεις για την επεξεργασία δεδομένων, για την πρόληψη της απάτης και την διαχείριση των κινδύνων. Είναι στόχοι που μπορούμε να επιδιώξουμε και αυτά προβλέπεται στα άρθρα για επεξεργασίες βάση συμφερόντων, ισορροπία συμφερόντων, ενώ θα κρατούμε ισορροπία με τα ενδιαφερόμενα άτομα. Γενικά για την Κομισιό η μείωση του φόρτου του διοικητικού είναι κάτι το σημαντικό και είμαστε στη διάθεσή σας για να εργαστούμε με τον συννομοθέτη για το στόχο αυτό ενώ θα κρατούμε τον, το επίπεδο προστασίας που δεν είναι προσδιορισμένη. Αναφέρομαι τους mitigating factors και σε αυτούς τους παράγοντες ε, η πρόταση λέει in particular δηλαδή ιδιαίτερα, αλλά όχι μόνο αυτά τα στοιχεία που αναφέρονται στον κατάλογο και όσον αφορά στα ποσά που αναφέρονται, είναι μέγιστα ποσά. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία που, θα, μπορούν να ληφθούν υπόψη και κάθε αρχή προστασίας δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα κριτήρια, θα εξετάσει κάθε περίπτωση ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της. Προτού αναφερθώ σε άλλα σημεία, θα ήθελα σύντομα να αναφερθώ στα σχέδια συμβιβαστικών τροπολογιών, που είναι ο ρόλος που θα ανατεθεί στο Open Protection Data Board, στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων το ανοιχτό. Το Συμβούλιο αυτό θα έχει αρμοδιότητα γνωμοδότητης, ενώ οι εθνικές αρχές έχουν αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων επειδή το board δεν έχει την αρμοδιότητα την νομική αυτή καθεαυτή και δεν υπάρχει μηχανισμός προσφυγής για, για, για αποφάσεις του board. Οι αποφάσεις του board είναι, αν θέλετε, γνωμοδοτήσεις. Για να απαντήσω ε, στις ειδικέ ερωτήσεις ε, της εισηγήτριας σχετικά με την διάταξη για το profiling. Ε, αντίθετα με τον κλασικό καθεστώς που είναι ένα καθεστώς ε, πλαισιωμένης ελευθερίας, το profiling ή ε, βασίζεται σε απαγόρευση με ιδιαίτερες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις. Δεν υπάρχει απόλυτη απαγόρευση επεξεργασίας δεδομένων, είναι ένα καθεστώς που βασίζεται σε ρητές εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις. Έχουμε διάφορα σημεία που μπορούμε να αναφέρουμε σε σχέση με το θέμα αυτό. Να υπενθυμίσω πρώτα απ' όλα ότι το καθεστώς για το profiling είναι η ε, συνέχεια του σημερινού καθεστώτος. Οι δραστηριότητες που επιτρεπόντουσαν από την υφιστάμενη οδηγία δεν απαγορεύονται από το νέο καθεστώς. Γιατί μιλάμε, μιλάμε για μέτρα που έχουν συνέπειες νομικές ή μέτρα που επηρεάζουν με σημαντικό τρόπο ένα άτομο. Δεν είναι κάθε δραστηριότητα profiling. Είναι ορισμένες δραστηριότητες που έχουν συνέπεια νομική για το άτομο ή το επηρεάζουν με σημαντικό τρόπο. Άλλο στοιχείο που βρίσκουμε στην πρόταση είναι ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Αν έχετε μια παρέμβαση ανθρώπινη ταυτόχρονα με την δραστηριότητα του υπολογιστή, δεν έχουμε ένα ε, μέτρο που είναι αυτοματοποιημένο επεξεργασίας. Έχουμε δραστηριότητες που βασίζονται αποκλειστικά σε επεξεργασία. Θα πρέπει να αξιολογούν ορισμένες απόψεις που σχετίζονται με ένα άτομο, να αναλύουν και να προβλέπουν την επίδοση στον τρόπο εργασίας, ε, τις προτιμήσεις, ε, την υγεία, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά του. Πότε ε, ε, εγκρίνεται το profiling. Αυτό το profiling επιτρέπεται όταν η ισορροπία ανάμεσα στο profiling και το άτομο λαμβάνεται αρκετά υπόψη. Μέσα στο πλαίσιο λοιπόν το συμβατικό είτε η διαπραγμάτευση προ συμβατική εκτέλεση κατόπιν ετήσεως ατόμου ή της εγγύησης για να υπάρξει παρέμβαση ανθρώπινη. Παραδείγματος χάρη σε σχέση με τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν ως ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αυτό γίνεται κατόπιν αιτήματος του ενδιαφορεμένου ατόμου. Μπορεί λοιπόν να μπει σε αυτή την κατηγορία. Αυτό το παράδειγμα, το marketing, ένα άλλο παράδειγμα που αναφέρθηκε, το marketing ε, δεν έχει συνέπειες νομικές για το άτομο ή δεν επηρεάζει το άτομο με ε, τρόπο σημαντικό. Η περίπτωση λοιπόν του παραδοσιακού marketing ε, δεν επηρεάζεται από αυτές τις διατάξεις. Να προσθέσουμε επίσης ότι το profiling επιτρέπεται είτε βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου είτε βάσει του εθνικού δικαίου που περιλαμβάνει κατάλληλες εγγυήσεις και οι διατάξεις για το profiling ενισχύονται από το άρθρο 21 ε, που παραπέμπει οριζόντια στην δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να παρεκκλίνουν από αυτές τις διατάξεις, κυρίως για λόγους δημοσίου συμφέροντος ε, για λόγους οικονομικούς, χρηματοοικονομικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κρατών μελών για συμφέροντα δημοσιονομικά, φορολογικά και προστασίας της σταθερότητας των αγορών. Άλλη δυνατότητα για να επιτραπεί το profiling είναι με τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ατόμου και με τις κατάλληλες εγγύησεις. Και επιμένω πάνω σε αυτό διότι η συμβατική αναγκαιότητα είναι μία δυνατότητα και το profiling είναι μία άλλη δυνατότητα. Υπάρχει μια ειδική διάταξη σύμφωνα με την οποία όχι αυτοματοποιημένο profiling και πάντοτε ε, μέσα στο πλαίσιο που είπαμε για τη συνέπεια την νομική ή την επίδραση την σημαντική για δεδομένα ε, ευαίσθητα για την εθνοτική ε, προέλευση, την φιλή κλπ. Έχουμε το γεγονός ότι ως προς το δικαίωμα πρόσβαση στα πλαίσια του άρθρου 20 υπάρχει μια πληροφορία που θα πρέπει να δίδεται για την, το νόημα και τις συνέπειες του profiling και στο άρθρο 20 υπάρχει μια αναφορά σε μια άλλη πληροφορία που θα δίδεται στα ενδιαφερόμενα άτομα. Το άλλο σημείο που αναφέρθηκε για τις μικρόμεσες επιχειρήσεις και το θέμα του κατοφλιού. Το κατόφλι που προτάθηκε από την Κομισιό είναι κάτι που βρίσκουμε σε άλλες πολιτικές. Το κατόφλι των 250 ατόμων αντιστοιχεί στον ορισμό των μικρόμεσαίων επιχειρήσεων στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, πράγμα που εξασφαλίζει μια συνακτικότητα σε σχέση με το κατόφλι αυτό. Γιατί προτείναμε ένα κατόφλι για να απλουστεύσουμε τη ζωή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βεβαίως σε αυτή την περίπτωση η μικρομεσαία απαλλάσσεται από φόρτο διοικητικό, δεν πρέπει να κάνει απολογισμό της ε, κατάστασής της, εκτός αν η βασική της δραστηριότητα είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Έχουμε λοιπόν εδώ ως σκοπό να μειώσουμε τον φόρτο των διοικητικών, να έχουμε ασφάλεια νομική και ένα κριτήριο ομοιόμορφο που εφαρμόζεται οριζόντια. Όσον αφορά στο θέμα των ανηλίκων, Σημεριζόμαστε τα όσα είπαν προλαλήσοντας ότι δηλαδή το είχαμε πει και στην προηγούμενη συνεδρίαση διαλέξαμε ένα κριτήριο που βασίζεται σε σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών η ηλικία των 18 ετών που είναι μια κοινή αναφορά, σημείο αναφορά όλων των κρατών μελών. Ίσως να σταματήσω εδώ για να μην παρατείνω κατά πολύ τη συζήτηση, αλλά να τονίσω ότι είμαστε στη διάθεσή σας, γιατί υπάρχουν πολλά άλλα σημεία για τα οποία θα μπορούσα να σχολιάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, για αυτές τις ε, πλήρεις ε, απαντήσεις, τις πολύ χρήσιμες που θα μας επιτρέψουν να ασχοληθούμε με τα θέματα στα οποία αναφερθήκατε. Είναι ένα θέμα αρκετά σημαντικό και αρκετά περίπλοκο. Κυρία Κόμη, θέλετε ίσως να συνοψίσετε ή να προσθέσετε ορισμένα σημεία. Ναι, πολύ σύντομα. Ως αφορά τις συναντήσεις μας και εγώ συμφωνώ. Στην, στο Στρασβούργο προσπαθήσαμε να το οργανώσουμε την Τετάρτη. Τελικά αυτό δεν κατέστη δυνατό γιατί δεν μπορούσαν να έρθουν κάποιοι βουλευτές ή κάποιοι υπάλληλοι. Αλλά αυτή είναι η καλύτερη λύση στις περιπτώσεις αυτές. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια απάντηση σε αυτά τα πολύ λεπτά ζητήματα και μόνο από τη διαπροσωπική μας συζήτηση μπορεί να γίνει αυτό. Γι' αυτό και χρειάζεται μια συνάντηση. Όταν λοιπόν επανέλθουμε τον Γενάρη να συναντηθούμε για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Για να μην χάνουμε χρόνο, εγώ έχω αποστείλει ε, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις τροπολογίες έτσι ώστε να έχετε να είναι εις γνώση σας το γενικό πλαίσιο. Αν θέλετε να προσθέσετε άλλα σημεία, άλλα στοιχεία. Να το κάνετε αυτό πριν από την πρώτη μας συνάντηση τον ε, Ιανουάριο ε, και έτσι να μπορέσουμε <clears throat> να τα εντάξουμε. Γιατί η ψηφοφορία είναι στις 24. Στις 23 η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ παρουσιάζει το σχέδιο ε, πρέπει να δούμε τι θα παρουσιάσουν και η Επιτροπή αυτή. Υπάρχουν, ε, είναι, έχουμε κάποια μειονεκτήματα, δεν έχουμε κοινή προσέγγιση με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ε, σταματώ εδώ το σχολιασμό μου. Σημείωσα όσα είπατε και θα μιλήσουμε. Στο μεταξύ σας, ευχα... σας εύχομαι καλή πρωτοχρονιά και καλά Χριστούγεννα. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα είναι καλή ιδέα να υπάρξει αυτή η συνάντηση τον Ιανουάριο, γιατί θέλω να είμαστε καλά προετοιμασμένοι για την ψηφοφορία και να δώσουμε την ευκαιρία στους συναδέλφους ε, να παρακολουθήσουν και τις, ε, ε, τα τεκτενόμενα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία και εδώ ολοκληρώνουμε κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω ότι αύριο στις 9 ξαναρχίζουμε. Έχουμε πάρα πολλές ψηφοφορίες, πια πολύ πολύ άσχολη ημέρα αύριο. Μην ξεχάσετε να φέρετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες για την ψηφοφορία. Επίσης θα, λάβουμε και θα βγάλουμε και μια συλλογική φωτογραφία. Θα υπάρχει ένας φωτογράφος εδώ θα βγάλουμε τη φωτογραφία μας που θα την έχουν στη διάθεσή τους όλοι για να μπορούν να την κάνουν και χριστουγεννιάτικο δώρο. Ε, θα μιλήσουμε λοιπόν εδώ, θα θέσουμε τις βάσεις για τον τριμερή διάλογο. Για... Ε, εύχομαι και πάλι καλά γενέθλια και χρόνια πολλά εδώ στον ε, συνάδελφο. Θα σας δω αύριο.